<coughs> Καλημέρα σας. Παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας. Θα αρχίσουμε την συνάντηση αυτή. Αυτή τη τόσο σημαντική, ιδιαίτερη μέρα που γιορτάζει την Διεθνή Μέρα της Γυναίκας του 2012. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τους συμμετέχοντες ότι μπορείτε να ακούσετε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. χάρη, το 11 ξέρω είναι σουηδικά. Μπορείτε να βρείτε λοιπόν σε ποιο κανάλι θα περάσει η σας γλώσσα, ελληνικά κάνει στο 7. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπορώ να σας παρουσιάσω τον νέο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Μάρτιν Σούλς. Παρακαλώ κύριε πρόεδρε, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Κούσταυσον. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω εγκαρδιότατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Διεθνή ημέρα της Γυναίκας είναι μια πολύ σημαντική μέρα εργασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια μέρα σημαντικών συζητήσεων μια ημέρα στην οποία αποστέλλεται ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα κάθε χρόνο από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε περήφανοι που η συζήτηση για την ισότητα των φύλων προωθείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια έντονα και με έντονε ε, διαμάχες και στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου και με άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, κρατών μελών. Προωθούμε τις σχέσεις μας ε, και με την ε, κοινωνία των πολιτών, συνδικαλιστικά κινήματα, πολιτιστικά κινήματα κλπ. Πάντα οι συνάδελφοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούσαν επαρκούς αυτούς ότι ήταν οι ηγέτες του κινήματος για την ισότητα των φίλων. Και ως πρόεδρος του σώματος θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε πρόεδρε και τους συναδέλφους σας για το έργο που επιτελείτε εδώ στη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Εργάζεστε ακούραστα ε, και η κυρίες και κύριοι που είναι τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών και ο κύριος Γκούσταυσον ως πρόεδρος ιδιαίτερα είναι ιδιαίτερα ισχυροί και μαχητικοί εκπρόσωποι του σώματος. Σας ευχαριστώ πολύ για την οργάνωση αυτής της διάσκεψης. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο Edit Power <coughs> που κάθεται εδώ εκ δεξιών μου. Η κυρία Μπάουρ είναι η συγγήτρια του σώματος για το θέμα της χρονιάς, όπως το έχουμε επιλέξει. Δηλαδή, ε, ίδιος μισθός για ίδια εργασία. Η συζήτηση αυτή για την ισοτιμία στην εργασία είναι κάτι που θεωρώ και εγώ, αλλά και που η πλειοψηφία του σώματος θεωρούν ότι είναι ένα κεντρικό θέμα στην δημιουργία κοινωνικής δικαιοσύνης ε, στην Ήπειρό μας. Προσωπικά για μένα, και το λέω εγώ ο άντρας και σύζυγος προσωπικά για μένα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και τις μεγαλύτερες ντροπέ θα έλεγα. Μια ντροπή είναι ότι για ίδια εργασία δεν πληρώνεται ο ίδιος μισθός. Η αρχή αυτή είναι μια τέτοια ταπείνωση εκείνων που εισπράττουν λιγότερα των γυναικών δηλαδή κυρίως, που καμιά φορά δεν βρίσκω λόγια για να μπορέσω να περιγράψω αυτή την ανισότητα. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που αυτό είναι το θέμα το φετινό. Ίσθιος μισθός για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα συζητήσετε αυτό το θέμα σήμερα με την κυρία Μπάουερ. δεν είναι κάτι που απλώς πρέπει να υποστηριχθεί, αλλά είναι μία από τις κύριες προκλήσεις και γι' αυτό είμαι ευγνώμων που είναι στο επίκεντρο των συζητήσεών σας τη σήμερα. Την περασμένη εβδομάδα είχα πάει στην Ελλάδα, κυρίε και κύριοι. Και θα επισκεφτώ και άλλες χώρες τη Ευρωπαϊκή Ένωση τι επόμενες εβδομάδε και του επόμενου μήνε. Ιδίω στις χώρε στις οποίε η οικονομική κρίση και η χρηματοπιστική κρίση πλήττει ε, τους πληθυσμούς και είδα την περασμένη εβδομάδα στην Ελλάδα ποιους πλήττει η κρίση αυτή κυρίως, τις γυναίκες και τους νέους. Η άνηση μεταχείριση των δύο φύλων σε περιπτώσεις κρίσης γίνεται ακόμα πιο εμφανής, χτυπάει πιο άσχημα. Και επιτρέψτε μου, ε, παρόλο που μιλάω σήμερα στην ημέρα των γυναικών υπέρ της ε, ισότητας, θα ήθελα να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι ντροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πιο πλούσια οικονομική ζώνη του κόσμου, χώρες που έχουν την πιο καλά εκπαιδευμένη ίσως νεολαία όλου του κόσμου. Νέους άντρες, νέες γυναίκες που υποφέρουν από ένα επίπεδο ενεργείας πάνω από το 50% δραματικό. Ακόμη πιο δραματικό για μένα είναι ότι πολλοί από αυτούς τους νέους, άντρες και γυναίκες, με τους οποίους μίλησα, δεν θεωρούν ότι είναι μηνύμα ελπίδας η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η πηγή των προβλημάτων τους. Και αυτό ισχύει και για πολλές γυναίκες που δικαίως θεωρούνται ότι διχανούν χάνουν άνησης, άδικης μεταχείρισης και ζητούν από μας, από την Ευρώπη, να πετύχουμε την ισότητα των φύλων και να εξαλείψουμε τις κοινωνικές ανισότητες και ότι θα πρέπει τα θέματα αυτά να είναι τα κεντρικά θέματα με τα οποία θα ασχολείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μπορώ να το καταλάβω αυτό. Όταν η κρίση πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες και όταν μεταξύ των νέων υπάρχει τόσο υψηλό επίπεδο ανεργίας, και το επίπεδο των μη απασχολουμένων νεαρών γυναικών είναι ακόμα υψηλότερο από το μη απασχολουμένων νεαρών ανδρών. Δηλαδή, σε, περι... σε εποχές κρίσης χτυπάει ακόμα περισσότερο αυτή η κοινωνική ανισότητα και η ανισότητα των φίλων. Και γι' αυτό είμαστε ακόμα περισσότερο υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τις οποίες θα συζητήσετε σήμερα όχι μόνο τις πρωτοβουλίες που υιοθετεί η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο για να διορθωθούν κάποια αριθμικά στοιχεία. Μου είπαν οι, ε, συνεργάτες μου σήμερα ποια είναι τα ακριβή στοιχεία που είναι φοβερά. 60% εκείνων που έχουν ε, δίπλωμα ε, πανεπιστημίου στην Ευρώπη είναι γυναίκες. Το 12,4% των γυναικών αυτών είναι στις διευθυντικές επιτροπές ε, μεγάλων επιχειρήσεων. σκανδαλώδες ήδη. Και 3,2% μόνο προέδρων των ε, επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι γυναίκες και 60% ξανατονίζω έχουν δίπλωμα πανεπιστημίου. Δεν χρειάζεται νομίζω να προσθέσω κανένα σχόλιο. Είναι εύγλωτα τα στοιχεία αυτά. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια πρωτοβουλία όπως εκείνο που υιοθετήθηκε υπό την αιγίδα της Vivian ε, Redding. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι νομικές, ε, νομοθετικές προϋποθέσεις για να αντιστρεφτεί ο κατάλογος αυτός. Κοίταξα τον κατάλογο των επισκεφτών που ήρθαν εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ. Τα θέματα που θα συζητήσατε, περιορισμό της βίας κατά των γυναικών, προστασία της μητρότητας, Ε, στην επίχρηματοδότηση αυτών των μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των κρατών μελών αλλά και μέσω της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στα πλαίσια των ε, συζητήσεων μας για τον προπολογισμό. Αυτά είναι κεντρικά θέματα. Ε, θα με απασχολούσαν και εμένα ως πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας εύχομαι για το μακρύ αυτό κατάλογο θεμάτων που θα σας απασχολήσουν σήμερα κάθε επιτυχία και ελπίζω να έχετε επικοδομητικές και αντιφατικές συζητήσεις, γιατί στην αντίφαση βασίζεται και η πρόοδος. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ο διάλογος μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι παρόντα εδώ και των επισκεπτών από τις διάφορες ε, κοινωνικο-οικονομικές, πολιτιστικές ομάδες που έχουν έρθει. Σας εύχομαι, λέω, να έχετε σήμερα μια επιτυχή ημέρα και συμβολικά επιτυχή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία για την εργασία σας. Και τελειώντα. θα ήθελα να εκφράσω μία παράκληση. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, είναι ένα θεσμό αν θέλετε, που, πώς να σα το πω τώρα, θα πρέπει να είχε την άδεια για την άσκηση κάποιου ε, επαγγέλματος εδώ, ε, πηγαίνω από εδώ εκεί συνεχώς, ε, μεταβιβάζομαι από τον ένα τόπο στον άλλο, από μια χώρα στην άλλη, στον, στην άλλη. Αν δεν μείνω εδώ κατά διάρκεια ε, της εργασίας σας, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχω διάφορες ε, άλλες υποχρεώσεις σήμερα. Μην θεωρήσετε ότι είμαι αγενής εάν φύγω τώρα, ολοκληρώνοντα την ομιλία μου. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Uh, uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρήκατε χρόνο να είστε εδώ. Ήταν ε, πάρα πολύ καλό το ότι ήρθατε, καλή διαφήμιση και δείχνει πόσο σημαντικό είναι το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα. Χαιρόμαστε που ήσασταν εδώ, έστω και για λίγο γνωρίζουμε πόσο βεβαρημένο είναι το πρόγραμμά σας. Επομένως και αυτή η λίγη ώρα που ήσασταν εδώ είναι σημαντική για εμάς. Σας ευχαριστούμε. Okay. Once again, good morning everybody. Να σας καλημερίσω για μια ακόμη φορά. Να καλωσορίσω όλους ιδιαίτερως 25 ε, μέλη από Εθνικά Κοινοβούλια 19 ε, βουλών άνω και κάτω από 16 κράτη-μέλη, των οποίων και υποψήφια ε, δύο είναι τα, πέντε είναι τα μέλη από δύο υποψήφιες χώρες. Να καλωσορίσω και όσους και όσες ευρωβουλευτές, ευρωβουλευτές είναι εδώ και να καλωσορίσω ε, τους πρώτους ομιλητές μας, Ένοτ Στάρκ και Πάρεντ Τυριό. Αλλά βέβαια να καλωσορίσω και όλους όσους συμμετέχουν ε, στις εργασίες μας είστε καλοδεχούμενοι σε αυτή την πολύ σημαντική συνεδρίαση. Αποτελεί παράδοση εδώ και χρόνια ε, και για μια ακόμη χρονιά έχουμε αυτή την εκδήλωση για να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις επ' ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας ε, των γυναικών που για πρώτη φορά γιορτάστηκε το 1911 πάνω από ένα εκατομμύριο γυναίκες και άνδρες ε, γιόρτασαν ε, στις ε, διάφορες εκδηλώσεις που είχαν διοργανωθεί την Διεθνή μέρα των γυναικών. Στόχος ήταν η μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών, η κατάργηση των διακρίσεων. Η Βιρτζίνια Γούλφ είχε μιλήσει για το πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες να έχουν το δικό τους χώρο. και μάλιστα ε, όχι μόνο χώρα αλλά και χρήματα δικά τους. Αυτή ήταν μια αλήθεια τότε, αλλά εξακολουθεί να είναι και σήμερα, γιατί η οικονομική ανεξαρτησία, αυτονομία των γυναικών είναι κεντρική σημασία για να είναι πιο ισότιμες οι σχέσεις των δύο φίλων στην κοινωνία. Βέβαια δεν είναι το μόνο, αλλά σίγουρα είναι ένα κομβικό στοιχείο. Εξού και η Επιτροπή Γυναικών θεωρεί ότι πρέπει για τη Διεθνή ημέρα ε, της γυναίκας του 2012 κεντρικό θέμα να είναι η ίση αμοιβή για ίση εργασία. Η εστίαση στα οικονομικά ζητήματα και την οικονομική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένα θέμα σημαντικό ε, σε μια εποχή όπου πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν οικονομική ύφεση και αυξανόμενη είναι η ε, ανισότητα που παρατηρείται μεταξύ ανδρών και γυναικών και στον τομέα των αμοιβών. Αυτό είναι ένα απαράδεκτο. Είναι μια μεγάλη αδικία σήμερα στην Ευρώπη να υπάρχουν διαφορετικές αμοιβέ για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα μαζί με τους διακεκριμένους μας προσκεκλημένους θα στείλουμε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι πρέπει να αναλυφθεί δράση για να καθιερωθούν ίσες αμοιβέ, να καταργηθούν οι διακρίσεις στις αμοιβέ. Θα ακούσουμε λοιπόν το πρώτο πάνελ. Οι ομιλήτρες θα μας εκθέσουν την άποψή τους, θα μας πούν ε, πώς επηρεάζουν αυτές οι ανισότητες ε, στους μισθούς και εν συνεχεία θα έχουμε ένα δεύτερο πάνελ όπου θα ακούσουμε εθνικέ εμπειρίε από τα διάφορα εθνικά κοινοβούλια, βέβαια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έχουμε και μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για το πώ θα συρρυκνώσουμε αυτό το χάσμα τη διαφορετική αμοιβή ανδρών και γυναικών. Και θα ακολουθήσει εν συνεχεία το τρίτο πάνελ, στη διάρκεια του οποίου θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τι μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των διαφορετικών αμοιβών αδρών και γυναικών. Θα ακούσουμε την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ηθαγένειας, την κυρία Ρέντινγκ που θα είναι εδώ. Θα είναι επίσης και ο κύριος ε, Μπαγής, εδώ, ο υπουργό. Ε, ε, ε, των ευρωπαϊκών υποθέσεων και βασικός διαπραγματευτής από την Τουρκία. Ενώ μέλος του πάνελ θα είναι και η κυρία Edith Power που είναι μέλος Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και τη Μισότητα των Φύλων και η οποία είναι και η συγγήτρια της έκθεσης που έχει τον τίτλο «Εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβή για άνδρες και γυναίκες εργαζομένους ε, που εργάζονται μάλλον για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η κυρία Μπάουερ, λοιπόν, στο τρίτο πάνελ θα μας παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσής της και τους βασικούς του στόχους. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε εμπειρίε και βέλτιστες πρακτικέ τις οποίε θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στην έκθεση αυτή, η οποία θα ψηφιστεί στη συνεδρίαση τη Επιτροπή ε, για την Ήπειρο τη Νίκας τον Απρίλιο. Είμαι βέβαιο ότι θα είναι αποδοτική, πλούσια η συζήτηση, θα μα δώσει ιδέε και θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τι ιδέε αυτέ στην πράξη, στην ε, πραγματικότητα τη διαφορετική τη κάθε χώρα πριν δώσω το λόγο στους ομιλήτρους του πρώτου πάντα, να σας δώσω και κάποιες πρακτικές πληροφορίες. Υπάρχει ένα έντυπο συμμετοχή για τους βουλευτές. Το έχετε στο γραφείο επάνω, στα έδρανά σας. Και μπορείτε να γραφείτε για χρόνο αγόρευσης ή να στραφείτε στους κλητήρες, ε, αν δεν έχετε αυτό το χαρτί. Θα έχουμε λοιπόν τρία μέρη στη συζήτηση. Το πρώτο έχει ως ε, τίτλο την ε, κατάτμιση της ε, αγοράς εργασίας ως παράγοντα ανισότητας. Το δεύτερο τμήμα έχει ως στόχο το, τη συρρήκνωση, ως θέμα μάλλον τη συρρήκνωση του χάσματος των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και το τρίτο είναι το πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να στηρίξουν ε, τα, την αντιμετώπιση της, ε, του χάσματος αυτού. Μπορείτε να λάβετε το λόγο για ένα ή για περισσότερα μέλη, μέρη. Τρία λεπτά είναι ο χρόνος αγόρευσης για τους βουλευτές, για τον καθένα βουλευτή. Θέλουμε να επιτρέψουμε να τον περισσότερους να λάβουν το λόγο. Επίσης, άλλοι προσκεκλημένοι που δεν είναι βουλευτές θα έχουν ένα λεπτό χρόνο αγόρευση στη διάθεσή τους ο καθένας. Επομένως, χωρίς να χρονοτριβήσουμε άλλο, περνούμε στο πρώτο πάνελ. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στην κυρία Κάριν Ένοτ, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. Παρακαλώ. Καλημέρα σας, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ και να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας της γυναίκας της 8 Μαρτίου και να ευχηθώ ε, να έχουμε όλοι καλή μέρα με τις ε, εορτάζουσες. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που με προσκάλεσε να συμμετάσχω σε αυτό το πάνελ για την καταμερισμό της, ομάδα, της αγοράς εργασίας ως στοιχείο διάκρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή, αυτός ο κατακαιρματισμός ε, έχει παραμείνει αμύωτος στα τελευταία 15 χρόνια. Δυστυχώς με εντυπωσιάζει αρνητικά αυτό το σύνθημα που ακούμε ίση αμοιβή για ίδια παρόμοια εργασία. Γιατί διαπιστώνουμε ακόμη ότι υπάρχουν διαφορές. Η TUC ενδιαφέρεται περισσότερο για την πραγματική υλοποίηση αυτού του συνθήματος. Για μας ε, είναι πιο ευστοχό το σύνθημα ίση εργασία για παρόμοια αξίες δουλειά. Βέβαια έχουμε ταυτόχρονα και την κρίση και η ίση αμοιβή βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας γιατί σήμερα αμέσως της κρίσης η ίση αμοιβή ε, για ίση εργασία είναι σημαντικότερη από, από ποτέ. Βέβαια ο, ο κατακαιρματισμός της αγοράς εργασίας διαπιστώνεται και οριζόντια και εγκάρσια σε διάφορους κλάδους και σε διάφορα επαγγέλματα. Δηλαδή, οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετικές ε, συνήθως ε, δουλειές. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει έξι επαγγέλματα με την μεγαλύτερη συμμετοχή. Ε, στα μαγαζιά πολίτριες είναι η θέση όπου απασχολούνται περισσότερο, απασχολούν περισσότερο οι γυναίκες. Δεν νομίζω ότι έχουμε εδώ περισσότερο συμμετέχοντες. Βέβαια έχουμε και ε, υπαλλήλου, οι εργαζόμενες στα σπίτια. Ενώ στους άνδρες έχουμε περισσότερο οδηγούς, ε, δικαιωμένους εργαζόμενους και ε, προϊσταμένους ή διαχειριστές μικρών επιχειρήσεων. Στις ε, σκανδιναβικές χώρες η διαφορά στα επαγγέλματα... Ε, δίνει τις γυναίκες να επικρατούν στο δημόσιο, ενώ οι άνδρες περισσότερο απασχολούνται στον ιδιωτικό κλάδο. Αν δούμε την εγκάρσια ε, διαφορά από μόνωση, βλέπουμε ότι ε, οι γυναίκες έχουν χαμηλότερους μισθούς και δεν απασχολούνται σε διευθυντικές θέσεις. Και οι διαφορές μισθών εξαρτώνται από τα επαγγέλματα και τους διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Πάντως είναι γεγονός ότι οι άνδρες και οι γυναίκες εργάζονται σε διαφορετικά επίπεδα των κλάδων και οι γυναίκες ε, απασχολούνται στις ε, χαμηλότερες, ε, χαμηλότερα μηδόμενες θέσεις. Και ο κατακαιρματισμός αυτός της αγοράς εργασίας θεωρείται ως ο βασικότερος λόγος για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Γιατί λοιπόν οι γυναίκες εξακολουθούν να επικεντρώνονται σε ορισμένα επαγγέλματα μόνο, σε ορισμένες εργασίες. Γιατί τυπικά εμπόδια δεν υπάρχουν πια για τις γυναίκες και τους άντρες να διαλέξουν την ε, παιδεία, ε, τη μόρφωση και την ε, εργασία που επιθυμούν. Και μάλιστα οι γυναίκες έχουν και καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο συνήθως από ότι οι άνδρες. Βέβαια, για τις επιλογές λαμβάνονται υπόψη και τα ενδιαφέροντα του καθενό. Οι γυναίκε έχουν περισσότερα ενδιαφέροντα, αλλά δεν είναι αυτό ο μοναδικό λόγο για την ε, στεγανοποίηση ορισμένων επαγγελμάτων. Σίγουρα οι γυναίκε έχουν και οικογενειακέ υποχρεώσει, εργάζονται περισσότερο με την οικογένεια και του ε, και ασχολούνται με τα παιδιά, οπότε έχουν λιγότερε λιγότερες πιθανότητες για επιτυχημένη σταδιοδρομία. Υποχρεούνται να διαλέξουν επαγγέλματα που η μερική απασχόληση είναι αποδεκτή. Σε τέτοιου είδου καταστάσεις δεν θα ευνοηθούν οι γυναίκες να μειώσουν αυτό το μισθολογικό χάσμα που υπάρχει. Μία εξήγηση όμως θα μπορούσε να είναι ότι οι γυναίκες επιλέγουν την αμερική απασχόληση επειδή οι άνδρες ε, προτιμούν πραγματική απασχόληση, δουλειά για ανδρε δηλαδή μία πλήρη απασχόληση και μερικές φορές μάλιστα με υπερορίες. Η επιλογή της μερικής απασχόλησης μάλιστα δεν είναι πάντα ελεύθερη. Ε, μερικές φορές είναι η μοναδική επιλογή που έχουν οι γυναίκες. Θα έλεγα μάλιστα ότι μερική απασχόληση σε ένα κλάδο που δεσπόζεται από τις γυναίκες, σε ένα επάγγελμα, ε, συνδυάζεται με την κατανομή των ε, υποχρεώσεων στο σπίτι και της φροντίδας των παιδιών. Αν, κανένας, ε, αν κάποια γυναίκα έχει μερική απασχόληση, Δυστυχώ, οι προοπτικέ αντιδρομίε είναι πολύ μικρές, οπότε η έκθεση προς την ε, φτώχεια, οι προς ε, πολύ χαμηλέ συντάξει είναι μεγαλύτερη. Δυστυχώς ε, πολλές γυναίκες πολύ καθυστερημένα το αντιλαμβάνονται αυτό, όταν είναι πια πολύ αργά για να αντιστρέψουν αυτή την πορεία. Υπάρχει όμως μία τάση ε, πολύ μορφωμένες γυναίκες ε, να εργάζονται λιγότερο σε θέση μερική απασχόλησης και αν επιλέγουν τη μερική απασχόληση θα το κάνουν για πολύ μικρότερη περίοδο. Βέβαια, είναι δύσκολο να γίνει μια τέτοια αξιολόγηση ε, και αυτό ιδιαίτερα στις χαμηλές, χαμηλά αμοιβόμενες θέσεις. Πάντως, πολλές φορές έχουμε ε, συστήματα αξιολόγηση που είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, ε, ακόμη και όταν χρησιμοποιούμε συστήματα αξιολόγηση τη εργασίας, ε, δύσκολα βρίσκουμε τα στοιχεία της αξιολόγησης ή δύσκολα βρίσκουμε συμφωνία για αναβάθμιση των μισθών στα κατάλληλα επίπεδα. Οπότε, τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις ε, θέσεις, πιο διευθυντικές ε, υψηλόβαθμες θέσεις. Περισσότερο εκεί απασχολούνται οι άνδρες, γιατί οι γυναίκες δύσκολα συνδυάζουν διευθυντικές θέσεις με τη φροντίδα των παιδιών ή την και του ζωή. Γι' αυτό είναι και πολύ πιο απρόθυμες ε, να κυνηγήσουν τέτοιες θέσεις. Είναι ένας λόγος αυτός επίσης για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Βέβαια, αυτή η στεγνοποίηση των ε, επαγγελμάτων και αυτό το μισθολογικό χάσμα μπορεί να βελτιωθεί με την ανίσχυση ε, του συστήματο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αλλά πιο σημαντική είναι η βούληση και η επιθυμία και των κοινωνικών εταίρων και των πολιτικών θεσμών να βρουν τι σωστέ λύσεις. Η πολιτική και οι θύνοντες θα πρέπει να βρουν τους σωστούς μηχανισμούς ε, για να επιτρέψουν την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας και την παραμονή τους. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν ε, συνεπείς και συνεκτικές πολιτικές, αναλαμβάνοντας ε, διάφορες ευθύνες και ε, επιδιώκοντα συμφωνία στην οδηγία για την άδεια μητρότητα. Επίση, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμφωνήσουν για την οδηγία του ωραρίου εργασία με διατάξει φιλικέ και προ την οικογενειακή ζωή. Βέβαια, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να επιδιώξουμε συνένεση και ελπίζω η συνένεση αυτή μεταξύ των ενδιαφερομένων να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Γιατί όλοι θέλουμε να υλοποιήσουμε το στόχο τη στρατηγική του 2020 και το στόχο για 75% απασχόληση και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Για να υλοποιηθεί όμως αυτός ο στόχος θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αντιληφθούν την ανάγκη μιας ισχυρής και συνεκτικής πολιτικής για το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, κάτι που σημαίνει καλύτερη φροντίδα των παιδιών, αλλά και καλύτερες οδηγίες για ρύθμιση, ε, μεταξύ, ε, ρύθμιση ε, της του συνδυασμού της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Φυσικά και ο ρόλος των θεσμικών οργάνων είναι πολύ σημαντικός για να φέρουν τα θέματα αυτά σε δημόσια συζήτηση και να ε, θεσπίσουν κοινοτικό δίκαιο και κοινοτικέ κατευθυντήριε γραμμέ. Αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ε, κεντρικό ρόλο να διαδραματίσουν, ζητώντα ε, νέα μέσα ισότητα φύλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζοντα με σωστό τρόπο την ήδη υπάρχουσα κοινοτική νομοθεσία. Νομίζω ότι η επένδυση στις γυναίκες και την οικογενειακή ζωή είναι μια αποδοτική επένδυση για τις γενικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στρατηγική του 2020. Σας εύχομαι λοιπόν καλή τύχη για αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Mrs. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ένοντ. Περνάμε στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Νιέτα Στάρκ, καθηγήτρια οικονομίας, οικονομικών από τη Σουηδία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ο εορτασμό της Διεθνού ημέρας ε, γυναικών συχνά όπως πρέπει είναι μια ημέρα αγανάκτησης αλλά και οδύνη για γυναίκες οι οποίες θανατώνονται, βιάζονται, κακοποιούνται σε ολόκληρο το χρόνο. Θύματα σεξουαλικής βίας, ε, ε, φτώχεια, στέρηση εξαθλίωση. Αλλά θα ήθελα να εκμεταλλευτώ σήμερα το πρωί την ευκαιρία που μα δίνεται για να χαιρετήσω και μια καθολική οικουμενική επιτυχία, αυτή που, που παρατηρείται στον τομέα της εκπαίδευσης τα τελευταία 50 χρόνια. Βλέπουμε μεγάλη αύξηση ε, των ε, μορφωτικών επιπέδων στην Ευρώπη, στον ΟΣΑ και ανά τον κόσμο. Η κοινωνία της γνώσης πραγματικά αυξάνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Μια μεγάλη πρόοδος συντελείται και πρέπει να την χαιρετήσουμε. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την αλληλεξάρτηση μεταξύ <clears throat> παιδείας και αγοράς εργασίας και έχουμε αυτό το στοιχείο του κατακαιρματισμού της κατάτμισης ε, της αγοράς. Ε, σήμερα, την εποχή της οικονομικής αναδιάρθρωσης, ίσως ε, βιώσουμε έναν φαύλο κύκλο διαχωρισμού, απομονωτισμού ή να δούμε αντιθέτως πρόοδο προς ένα μέλλον με μεγαλύτερη ισότητα. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες για δράση. Και βέβαια το σημαντικότερο είναι η μελλοντική οργάνωση των κοινωνιών μας και το πώς μπορούμε στο μέλλον να εξασφαλίσουμε ότι μεγάλα τμήματα της κοινωνίας μας θα μπορούν να λειτουργούν εύρυθμα στο μέλλον. Ότι θα έχουμε άτομα ανταγωνιστικά που θα μπορούν να αποδίδουν και να λειτουργούν ε, σε όλες τους τις ευθύνες τα καθήκοντά τους. Και επίσης πώς μπορούμε σε ατομικό επίπεδο να δώσουμε σε κάθε άντρα, σε κάθε γυναίκα δυνατότητες για εργασία και αμοιβόμενη και μη αμοιβόμενη Πώ πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ε, δεξιότητές τους για να τις πασαρμόσουμε στις ανάγκες. Να σας πω κάποια στοιχεία. Οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία ε, φοιτητών από φοιτών πανεπιστημίων σχεδόν σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Χρησιμοποιώ στατιστικά στοιχεία ε, από τον ΟΣΑ και όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για σήμερα, γιατί θα ήθελα να δώσω μια ευρύτερη, πιο διεθνή προοπτική. Οι γυναίκες επίσης στον τομέα της παιδείας, της υγείας ε, και της πρόνοιας ε, δεσπόζουν. Μιλάμε για βασικές ανάγκες βέβαια της κοινωνίας, αλλά και στις ανθρωπιστικές επιστήμες μεταξύ άλλων. Και νομική. επίσης οι άνδρες στη μηχανική, στις κατασκευές είναι αυτοί που εκπροσωπούνται περισσότερο, σπουδάζουν ε, μια ε, ευρεία κάμα οι γυναίκες ε, μαθημάτων, ευρύτερη από αυτή των ανδρών. Και αυτό το βλέπουμε να το αντικατοπτρίζεται και στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε όλους τους τομείς, βέβαια υποεκπροσωπούνται στην μηχανολογία ή στις κατασκευές, αλλά ενώ πριν από κάποιες δεκαετίες υπήρχε κυριαρχία των ανδρών σε τομείς όπως η νομική, το δίκαιο κτλ. Αυτό πλέον δεν ισχύει. <clears throat> τα ποσοστά αποφύτηση για τις γυναίκες στις χώρες του ΩΣΑ είναι πολύ ψηλότερα σε σχέση με τους νεαρούς άνδρες. 46% των νεαρών γυναικών έχουν ε, πλέον ένα ανώτερο τίτλο σπουδών σε σχέση με τους άνδρες, που το αντίστοιχο νούμερο είναι 31%. Άρα μιλάμε για 15 ποσοστιαίες μονάδες σε βάρος των ανδρών. Περισσότερες γυναίκες. Οι γυναίκες επίσης ε, εδώ και κάποιο καιρό ε, εκπαιδεύονται περισσότερο ε, και δεν μιλάμε μόνο για την υψηλοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για την, τον αλφαβητισμό σε χώρες όπως η Ναμίμπια, παραδείγματος χάρη, η Μποτσοάνα, η μάθηση στην Ανατολική Ασία, στη Λατινική Αμερική. Σε μεγαλύτερη ηλικία βλέπουμε οι γυναίκες περισσότερο να ενδιαφέρονται να σπουδάσουν. Οι γυναίκες πραγματικά αγαπούν ε, την εκπαίδευση. Μην ανησυχείτε όμως, τις, ε, ε, τα ανώτερα κλιμάκια στα πανεπιστήμια εξακολουθούν να βρίσκονται άνδρες. Θα ήθελα να σας πω Τώρα για την εκπαίδευση, για την, ε, θα το χωρίσω στο ατομικό και στο δημόσιο επίπεδο. Γιατί οι χώρε του ΩΣΑ χρησιμοποιούν ε, τα δημόσια ταμεία για να δουν ε, ποια είναι η δημόσια, ποιο είναι ο δημόσιο αντίκτυπο, ποια είναι τα ιδιωτικά κέρδη από την εκπαίδευση. Είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή για τα άτομα τα οποία πηγαίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή που σπουδάζουν σε ένα πανεπιστήμιο. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση φέρνει πολύ σημαντικές ανταμοιβέ σε πολύ μεγάλο αριθμό χωρών. Στις χώρες του ΩΣΑ μιλάμε για ευρία γκάμα χωρών. Περιλαμβάνεται και το Μεξικό για παράδειγμα. Ο εργασιακό βίος για έναν άντρα αποφέρει 175.000 δολάρια περισσότερο σε έναν άντρα που έχει σπουδάσει παρά σε έναν που δεν έχει σπουδάσει. Ενώ για τη γυναίκα η αντίστοιχη αμοιβή είναι 110.000. Άρα 65.000 ε, δολάρια λιγότερα. Για ποιο λόγο? Γιατί κερδίζουν περισσότερα οι άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, παρότι έχουν τα ίδια, τις ίδιες σπουδέ, είναι στο ίδιο επίπεδο σπουδών. Ποια είναι τώρα τα δημόσια κέρδη, τα δημόσια ωφέλη. Η απόδοση, η ε, επιστροφή, δηλαδή αν σκεφτούμε ε, τι απόδοση θα έχει να επενδύσει κανεί σε έναν άνδρα ή σε μια γυναίκα. Τα ποσά είναι 91.000 για του άνδρες, 55.000 για τι γυναίκε. Πάλι χαμηλότερα δηλαδή για τι γυναίκε. Ενώ απαιτούνται αντίστοιχα επίπεδα δεξιότητας. όλα αυτά ε, βλέπουμε εισοδήματα πιο υψηλά για τους άνδρες, αλλά βέβαια και περισσότερη φορολογία. Πληρώνουν πιο πολλού φόρου οι άνδρες. Τελικά, γιατί κανείς ε, να ε, προωθήσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση για τι γυναίκε. Καλύτερα σπουδάζουν μόνο οι άντρε στο πανεπιστήμιο και οι γυναίκε όχι. Φυσικά αυτό είναι μια αστεία, ένα αστείο συμπέρασμα. Υπάρχει και μια πιο λογική, ένα πιο λογικό συμπέρασμα. Έχουμε κάποια μελέτη του ΩΣΑ για το 2011. Δεν κάνει λοιπόν φυσικά τέτοια πρόταση ΩΣΑ. Τώρα, γιατί οι άντρε δεν στρέφονται πιο πολύ στην ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν του αρέσει να κερδίζουν χρήματα παραπάνω. Όχι, δεν είναι αυτή η απάντηση. Αν δεν έχουν ε, ένα πτυχίο τριτοβάθμια εκπαίδευση, κερδίζουν περισσότερα από τι γυναίκε παρόλα αυτά. Άρα καλύτερα τα καταφέρνουν οικονομικά από τι γυναίκε, ακόμη και αν δεν έχουν προχωρήσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μήπω δεν αρέσει στου άντρε ε, η μάθηση, δεν τους αρέσουν οι σπουδές. Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Οι γυναίκες είναι περισσότερες ε, στην τετοβάθμια εκπαίδευση από τους άνδρες. Γιατί? Γιατί αν δεν σπούδαζαν στην τετοβάθμια εκπαίδευση θα είχαν ακόμα λιγότερη αμοιβή σε σχέση με τους άνδρες. Αν δούμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί προβλέπουμε έλλειψη εργατικού δυναμικού. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προκαλέσω κάπως, ε, ε, έχει λίγο εγκαταλείψει τους άνδρες διότι η εκστρατεία, η καμπάνια στρέφεται μόνο ε, στο πώς θα προσελκύσει στις κατασκευές, στη τεχνολογία, στη μηχανολογία γυναίκες. Αν δεχτούμε, και εγώ δεν δέχομαι, αυτή την, ε, το διαχωρισμό, τη διάκριση ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εκπαίδευση, το λογικό θα ήταν να ενθαρρύνουμε περισσότερους άνδρες προς αυτή την κατεύθυνση που ούτω ή άλλως το συνηθίζουν. Βλέπουμε όμως ότι στρέφονται μακριά από την τριτοβάθμια εκπαίδευση οι άνδρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πλέον να ενθαρρύνει μόνο τις γυναίκες να προβούν σε ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές, για τις οποίες έχουν ήδη αποδειχθεί ικανότατες μέχρι τώρα. Θα ήταν λοιπόν το επικίνδυνο συμπέρασμα να πούμε ότι θα έπρεπε να αποθαρρύνουμε τις γυναίκες να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο. Αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος που έχει, σωστό, που έχει σωστά, στα σφρένα θα σκεφτόταν κάτι τέτοιο. Το σημαντικό λοιπόν δεν είναι μόνο να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να ασχοληθούν με νέους τομείς, αλλά να κινητοποιήσουμε τους άνδρες, να τους βγάλουμε από την άνεσή τους, ε, από τους τομείς στους οποίους νιώθουν άνετα, τις τεχνολογίες, τη μηχανολογία, τις κατασκευές. Και σας παρακαλώ όλους και όλες να σκεφτείτε τις αλλαγές που συντελούνται σήμερα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μάρτιν Σούλτ είπε κάποια πράγματα στην εισαγωγική του ομιλία. Τα μέτρα λιτότητα, τι αντίκτυπο θα έχουν σε βασικού τομεί απασχόληση για τι γυναίκε, δηλαδή η υγειονομική περίθαλψη, η ιατρική, ε, έρευνα, εκπαίδευση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποστραφούμε αυτό το οποίο έχω δει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια συζήτηση δηλαδή για τις γυναίκες μάλλον για ε, την υποψία που υπάρχει ότι μήπως υπερκαταναλώνουν οι γυναίκες ε, την ανώτερη, ανώτατη εκπαίδευση και δεν τη βλέπουν ως επένδυση αυτήν την ε, επένδυση των γυναικών. Μάλλον αυτήν την ε, ενασχόληση των γυναικών με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ουσιαστικά οι γυναίκες παίρνουν ίδιες την ευθύνη να επενδύσουν στη μεγαλύτερη εκπαίδευση. Οι γυναίκε λοιπόν θα πρέπει να είναι ε, ο νέος κανόνας, το νέο πρότυπο για περισσότερη εκπαίδευση. Άρα τώρα θα πρέπει να μας ανησυχούν οι άνδρες που δεν έχουν τις ίδιες επιδόσεις ή τέλος πάντων δεν έχουν τις επιδόσεις που θα θέλαμε εμείς ε, οι πολίτες να είχαν για την αποκτήση προσόντων, δεξιότητων, για τη μάθηση. Ίσως ε, είναι λίγο διαφορετική η απόχρωση που δίνω στη σημερινή συζήτηση. Αλλά ένας από τους λόγους για τους οποίους οι άνδρες δεν προχωρούν, ε, δεν ασχολούνται με νέους τομείς, είναι γιατί μένοντας εκεί που είναι κερδίζουν περισσότερα χρήματα. Οι γυναίκες έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν αλλάξει, έχουν προσαρμοστεί, μαθαίνουν νέα πράγματα. Αν πούμε ότι 3,2% των γυναικών βρίσκονται σε ανώτατα κλιμάκια σε ιδιωτικέ επιχειρήσεις, μπορούμε επίσης να πούμε ότι το 96,8% των θέσεων αυτό καταλαμβάνονται από άνδρες που δεν αποδίδουν ε, το ίδιο καλά με τις γυναίκες στην ανώτατη εκπαίδευση. Ας το έχουμε υπόψη μας αυτό. Άνδρες επίσης οι οποίοι περιμένουν αλλά και λαμβάνουν υψηλότερη αμοιβή σε σχέση με, την, ε, με τις γυναίκες για την ίδια, για το ίδιο επίπεδο δεξιοτήτων. Thank you. Σας ευχαριστούμε κυρία Στάρκ και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Παγαντηριών, εκπρόσωπο του Eurofound. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ θερμά ε, και την προλαλής, τις ε, για τις προκλητικές πραγματικά ομιλίες τους που θα δώσουν και τροφή στη συζήτηση. Επανέρχομαι στην παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασία, ε, στο εργατικό δυναμικό και θα ήθελα να αναπτύξω δύο ιδέες που έδειξαν οι προλαλήσαντες. Σε ό,τι αφορά τι επιλογέ που θα κάνουμε, τι είδο κοινωνία θέλουμε, τι είδο κόσμο θέλουμε, στον οποίο θα συμβιώνουν από κοινού άνδρε και γυναίκε. Επίση, θα ήθελα επαναφέρω αυτή την ιδέα της ε, απόδοσης των επενδύσεων, της επιστροφής ε, των επενδύσεων που ανέφερε η προλαλή σα. Ό,τι αφορά το διαχωρισμό των δύο φύλων ε, στην αγορά εργασίας. είναι γεγονό αυτός ο διαχωρισμός. Ακούσαμε τα αριθμητικά στοιχεία. Εγώ θα προσθέσω ακόμη μερικά για να τεκπηριώσω περισσότερο αυτή τη θέση με βάση μία απογραφή για τις εργασιακές ηθίκες σε 34 ευρωπαϊκές χώρες διαπιστώνουμε ότι 17% των ανδρών εργάζονται σε, ε, σε επαγγέλματα που εκπροσωπούνται και τα δύο φύλλα και 20% των γυναικών περίπου. Οπότε ε, οι περισσότεροι ε, δηλαδή εργαζόμενοι απασχολούνται σε επαγγέλματα που δεσπόζονται από ένα φύλλο μόνο. Λίγοι είναι οι εργαζόμενοι σε μεικτά επαγγέλματα αυτή το διαχωρισμό τον διαπιστώνουμε σε διάφορους κλάδους. Είπαμε στη μεταποίηση, στην ε, κατασκευή, ε, Επίσης ε, στις εταιρείες πολύ συχνά οι γυναίκες εργάζονται σε πιο μικρές επιχειρήσεις και ο διαχωρισμός αφορά και επαγγέλματα και οικονομικούς κλάδους και μεγέθη επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά το, τη γυάλινη οροφή κατά κάποιο τρόπο, είναι ενδιαφέρον και αυτό το φαινόμενο. Εξετάζοντας τα στοιχεία μας, διαπιστώνουμε αυτό το, τη γυάλινη οροφή, δηλαδή το ποσοστό α, όσων από το 1991 έχουν γυναίκα διευθύντρια. Μεταξύ του 1991 και σήμερα διαπιστώνουμε ότι η αύξηση ήταν 6%, ε, δηλαδή έχουμε 22% σήμερα. Αν θέλουμε να φτάσουμε το 45% ε, συμμετοχή των γυναικών, δηλαδή ε, όπως των γυναικών στην αγορά εργασίας, ή 50%, ίση συμμετοχή θα χρειαστούμε άλλα 40 έως 60 χρόνια για να εξασφαλίσουμε αυτό το ποσοστό, εκτός και αν φυσικά ε, σημειώσουμε πιο ραγδαία πρόοδο. Υπάρχει και αυτή η γυάλινη οροφή και δεν αφορά μόνο την χαμηλή συμμετοχή των γενικών σε διευθυντικές θέσεις, είναι ότι όταν είναι διευθύντρες οι γυναίκες, ε, ε, είναι διευθύντρες σε πολύ μικρότερες ομάδες, είναι προϊσταμένες σε πολύ μικρότερες ομάδες ή σε θέσεις μερικής απασχόλησης και εκεί υπάρχει δηλαδή ανισότητα. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι και το μισθολογικό χάσμα φυσικά. Οι περισσότερες ε, γυναίκες έχουν χαμηλότερες αποδοχές από τους άνδρες. Είναι 35% ε, σε όλες τις ε, ε, φάσεις της επαγγελματικής σταδιοδρομίας η διαφορά. Υπάρχει λοιπόν ο διαχωρισμός των δύο φύλων και είναι πολύμορφος και πολύ σύνθετος. Ένα άλλο σημαντικό κλάδο και μια άλλη σημαντική δραστηριότητα για μα είναι το θέμα τη ε, φροντίδα. Εκεί γίνεται ο συνδυασμό κυρίω από τι γυναίκε. Εκεί είναι που, θα που καλούνται να πραγματοποιήσουν κάποιε επιλογέ. Εμεί στην Ευρώπη αποφασίσαμε ότι 75% των ανδρών και των γυναικών θα, θα έχουν ε, μια απασχόληση και θα λάβουν ε, άδεια μεταποδοχών και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι θα πρέπει η φροντίδα να καλύπτεται σε αυτή την μεταποδοχών άδεια. Αυτό που έχουμε παραλείψει τελείω είναι οι συνέπειε αυτή τη επιλογή. Οι γυναίκε φέρουν τη μεγαλύτερη ε, ευθύνη για την φροντίδα των παιδιών. Θα πρέπει να δούμε τώρα αν αυτή η φροντίδα θα είναι μεταποδοχών ή άνευ αποδοχών και ποιο τμήμα της φροντίδας θα καλύπτεται από το μισθό. Μία άλλη επιλογή που θα πρέπει να κάνουμε είναι τι είδου ε, θέσεις απασχόλησης θα δημιουργήσουμε για αυτές τις ε, δραστηριότητες φροντίδας. Θα υποστηρίξουμε με κοινωνικό εισόδημα αυτές ε, τις δραστηριότητες. Για παράδειγμα, θα πούμε στις γυναίκε τώρα έχετε παιδιά, μπορείτε να λάβετε μία άδεια γονική και να επανέλθετε στην αγορά εργασία Ή θα πούμε βρείτε κάποιον άλλον που θα μεγαλώσει τα παιδιά σας, που θα τα φροντίσει. Ή θα οργανωθούμε συλλογικά και θα επιλέξουμε κάποιες προδιαγραφές. Αυτό είναι θέμα κοινωνικής επιλογής. Στην Ευρώπη έχουμε πολύ διαφορετικές συμπεριφορές για το θέμα αυτό και είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί και αυτό φυσικά θα επηρεάσει και τις απολαβές των γυναικών, την ποιότητα της εργασίας τους και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας και το είδος ε, συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Ποιες γυναίκες ε, θα κάνουν ε, αυτές τις επιλογές. Αυτό είναι σημαντικό ε, και για τους γονείς και για το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ε, ζωής και για τους εργαζόμενους. Έχουμε βέβαια τα κριτήρια της Βαρκελόνης και την δέσμευση ε, δημιουργίας υποδομών για τη φροντίδα των παιδιών. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, αλλά το θέμα δεν αφορά μόνο τη φροντίδα των παιδιών και την ανατροφή των παιδιών. Το θέμα αφορά και τις σχολικές υποδομές και το κατά πόσο το σχολείο, η διάρθρωση του σχολείου επιτρέπει τις γυναίκες ε, να συνεχίσουν τη δουλειά τους και τι γίνεται με παιδιά που έχουν ειδικέ ανάγκες ή ε, τι γίνεται με τη φροντίδα των ε, ηλικιωμένων. Ακόμη και όταν αποφασίσουν να μην αποκτήσουν παιδιά οι γυναίκες, πολλές φορές φροντίζουν τους ηλικιωμένους γονείς και είναι συνήθως οι γυναίκες που φροντίζουν τους ηλικιωμένους γονείς. Υπάρχουν διάφορες ε, δυνατότητες λοιπόν οργάνωσης, είναι θέμα επιλογής και επίσης ε, έχουμε διαφορετικά επίπεδα και ποιότητες εργασίας και αυτά είναι θέματα επιλογής που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ένα τρίτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η σχέση με το χρόνο. Όπως είπα και προηγουμένως, οι γυναίκες ε, θα έχουν μια δουλειά, ε, θα επιστρέψουν στο σπίτι τους για τις οικογενειακές υποχρεώσεις και πολλές φορές έχουν και δεύτερη ε, δουλειά για να αυξήσουν το εισόδημά τους. Πολλές φορές έχουμε γυναίκες ε, που απασχολούνται με μερική απασχόληση και εκεί βλέπουμε πόσο χρόνο αφιερώνουν στην κάθε δραστηριότητά τους. Είναι το, από το, το φαινόμενο σταχτοπούτας. Από τη στιγμή που αποκτά παιδιά η γυναίκα κάθε μέρα έχει και από όλες οικογενειακές υποχρεώσεις και ε, το επάγγελμά τη και μάλιστα ακόμη και όταν απασχολείται σε μερική απασχόληση, από τη στιγμή που έχει και παιδιά και προσθέσουμε την αμοιβόμενη και τη μη αμοιβόμενη εργασία, πάλι γυναίκε και με μερική απασχόληση εργάζονται πολύ περισσότερη ώρα από ό,τι άνδρε. Γιατί λοιπόν να μην αναλάβουν και άνδρες ένα τμήμα αυτών των ε, ε, μη αμοιβόμενων δραστηριοτήτων. Χρειάζονται όμω και κοινωνικέ υποδομές για κάτι τέτοιο, ίσω και κάποιοι κανονισμοί για το ωράριο εργασία, ε, για περιορισμό του ωραρίου εργασία, ώστε να είναι πιο εύκολο να συνδυάσουν οι γυναίκε ε, τι οικογενειακέ με τι επαγγελματικέ υποχρεώσει και ίσω να μην χρειάζεται καν να καταφύγουν στη μερική απασχόληση και άρα να μειώσουν το εισόδημά του με μια τέτοια μερική απασχόληση. Ε, είναι θέμα και συμπεριφορά φυσικά. Όταν ρωτούμε τους εργαζόμενους ε, αν πιστεύετε ότι η επαγγελματική σας ζωή συνδυάζεται με την ιδιωτική σας ζωή. Ε, οι περισσότερες γυναίκες απαντούν ότι είναι σε αυτός ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, γιατί οι γυναίκες και οι άνδρες ξεκινούν από διαφορετικό σημείο φετηρίας όταν ε, αποφασίζουν να εργαστούν. Οι άνδρες Ακόμη ε, μετά, όταν αποκτούν παιδιά, διαπιστώνουν πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Αλλά οι γυναίκε το ξέρουν εκ των προτέρων και προσπαθούν να προσαρμοστούν στι στις ε, καταστάσει. Προτιμούν φυσικά πιο ελαστικό ωράριο, αλλά γνωρίζουν α, ε, ότι είναι ικανέ να συνδυάσουν διάφορε δραστηριότητε μέσα στην ημέρα. Επίσης σημαντικό είναι και το θέμα της συμπεριφοράς της τάσης. Στην έρευνά μας έχουμε ένα δείκτη για μικρές ρυθμίσεις εντό συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Μέσα σε μία-δύο ώρες διάλειμμα, για παράδειγμα, πώς αντιμετωπίζουν έκτακτες περιστάσεις οι εργαζόμενοι. Διαπιστώσαμε στην έρευνά μας ότι είναι ευκολότερο για τους άνδρες να κάνουν κάτι τέτοιο από ό,τι για τις γυναίκες. Οπότε θα πρέπει να δούμε τη διάρκεια και ταυτόχρονα να δούμε και την ε, οργάνωση του ωραρίου εργασίας και τα δικαιώματα που έχουν, ε, αλλά και τη συμπεριφορά και τη στάση που έχουν άνδρες και γυναίκες. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θέξω είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει διαχωρισμό στην αγορά εργασία, είναι διαφορετική έκθεση και στου κινδύνου. Μία βασική πρόκληση είναι να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις ε, ασχολίες των γυναικών για να δούμε τι κίνδυνο ε, ελοχεύει σε κάθε ε, ασχολία και να υιοθετήσουμε προληπτικές δράσεις προκειμένου να αποσοβήσουμε αυτό το κίνδυνο. Είναι ενδιαφέρον για παράδειγμα να δούμε ότι όταν προσπαθούμε να καταμετρήσουμε έκθεση στην ε, μεταφορά ε, βαριών φορτίων είναι θέμα προβληματικό και πολλές γυναίκες το επισημαίνουν αυτό ε, αν στη δουλειά σας κουβαλάτε βαριά φορτία. Όταν αλλάζουμε όμως την ερώτηση και λέμε όταν κουβαλάτε ανθρώπους, παιδιά ας πούμε, όταν δεν έχουμε όρους φορτίου αλλά ανθρώπου, εκεί είναι περισσότεροι γυναίκες που κουβαλάνε από ότι οι άντρε. Υπάρχουν ε, διαφορές λοιπόν. Θέλουμε ποιοτικέ εργασίες για να ε, επιτρέψουμε και στους άνδρες και στις γυναίκες να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει πολυεπίπεδε πο... Ε, και πολυσύθετες δράσεις και αλλαγή της νοοτροπίας στην κοινωνία και η συγκεκριμένη επιλογή για το τι στόχους θέλουμε να υλοποιήσουμε. Και ας μην ξεχνούμε και την κρίση. Θα πρέπει παρά την κρίση να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πανετήριο. Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχω ήδη έναν κατάλογο μιλητών. Να ευχαριστήσω τις τρεις ομιλητριές μας. Ήταν πολύτιμη η συνεισφορά τους στη συζήτηση. Και τώρα θα ακούσουμε τα σχόλια του κοινού. Εν συνεχεία μπορείτε να απαντήσετε. Ερωτήσεις ή σχόλια λοιπόν από το κοινό, πρώτα απ' όλα από το ακροατήριο. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στην κυρία Μπάρμπαρα Μπόρις Σταμιέσκα από την Γερουσία, από την Πολωνία. Τρία λεπτά το πολύ έχετε στη διάθεσή σας κυρία μου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, μια και είμαι η πρώτη ομιλήτρια, να σα ζητήσω ένα μικρό μπόνου. Λοιπόν, αρχίζω. Ισχύει ο εργατικό κώδικα στην Πολωνία εξασφανίζει στου ε, εργαζόμενου δικαίωμα ίση αμοιβή για ίση εργασία ή για εφάμιλη εργασία. Και μάλιστα εδώ επαναλαμβάνεται το άρθρο 141 τη συνθήκη του Άμστερνταμ που επιβάλλει στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, την εξασφάλιση ε, της αρχής της ίσης ε, μεταχείρισης και ίσης, ίσου μισθού ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία. Την ίδια εργασία. Στα τέλη του 2010, ο αριθμός εργαζόμενων γυναικών στην Πολωνία ήταν 8.022.000, ενώ οι άνδρες 9.702.000. Παρά τις νομιμοθετικές διατάξεις, υπάρχουν διαφορές στις αμοιβέ ανδρών και γυναικών, που δυστυχώς είναι ακόμη αισθητές. Θα προσπαθήσω να μιλήσω συνοπτικά, να σας πω μόνο ότι στο δημόσιο η διαφορά ε, μισθού μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν 695 ζλότη ε, εις βάρος των γυναικών φυσικά, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η διαφορά αποδοχών ανδρών και γυναικών ενερχόταν σε περίπου 730. Μήπως θα μπορούσατε να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει ο Πρόεδρος, γιατί δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνείς. Επαναλαμβάνω ότι είναι σημαντική η, διαφορά αυτή των μισθών και μάλιστα πιο αισθητή είναι, είναι πιο σημαντικές αυτές οι διαφορές σε διευθυντικές θέσεις, σε υψηλόβαθμους υπαλλήλου. Ε, μάλιστα, οι διαφορέ αυτέ για του άνδρε ήταν 8.403 ζλότι, για τι γυναίκε 6.067 ζλότι. Δηλαδή, ε, βλέπουμε διαφορά 2.335 ζλότι μεταξύ ανδρών και γυναικών στου μισθού. Αυτέ οι ψηλόβαστες θέσεις, ενώ για τις τεχνικές ή για το μέσο προσωπικό οι διαφορές στους μισθού ήταν περίπου χίλια σλότη. Υπάρχουν κάποιε αλλαγέ βέβαια και βελτιώσεις, για παράδειγμα στο ποσοστό απασχόληση, στο μισθό, στο ωράριο εργασίας, στις διευθυντικέ θέσεις, στην κατανομή των υποχρεώσεων μεταξύ επαγγελματό και οικογένεια, έκθεση στη φτώχεια αλλά δεν έχουμε πολύ αισθητέ διαφορέ. Με βάση τι έρευνε που σα ανέφερα προηγουμένω, στι διευθυντικέ θέσει, οι γυναίκε ε, που εργάζονται στι μεγαλύτερε ε, ε, επιχειρήσεις κερδίζουν 5.700 ζλότι, ενώ οι άνδρες 7.000 ζλότι. Μάλιστα, οι γυναίκες σε θέση υπεύθυνου έργου ε, κερδίζουν 5.960 ζλότι, ενώ σε αντίστοιχη θέση οι άνδρες 8.000 ζλότι. δηλαδή 34% περισσότερο κερδίζουν οι άντρε. Ένας προϊστάμενος γραφείου ε, έχει μισθό 5.973 ζλότι ω άντρε, ενώ μια γυναίκα μόνο 4.410 ζλότι. Δηλαδή υπάρχει διαφορά 1.563 ζλότι ει βάρο των γυναικών. Τις μεγαλύτερες διαφορές ε, τις διαπιστώνουμε μεταξύ ανθρώπων που έχουν στοιχειώδη επαγγελματική κατάρτιση, όπου γυναίκες ε, κερδίζουν μόνο το 65% των ανδρικών μισθών. Το μισθολογικό χάσμα είναι πιο αισθητό στις γυναίκες άνω των 40 ετών. Εκεί είναι πολύ πιο αργός ο ρυθμός των προαγωγών και μάλιστα σε αυτή την ηλικία ε, οι γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερες διακοπές στην εργασία για τη φροντίδα των παιδιών και ιδιαίτερα ε, απασχολούνται οι γυναίκες στο δημόσιο, κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ πιο εκτεθειμένες σε απολύσεις εξαιτίας δημοσιονομικών περικοπών. Αυτά μάλιστα είναι τα στοιχεία της Κεντρικής ε, Στατιστικής Υπηρεσίας της Πολωνίας και παρόλο που πολλές μελέτες μας λένε ότι οι γυναίκες είναι ε, πιο μορφωμένες, καλύτερα οργανωμένες, αποκτούν γρηγορότερη πείρα στις διάφορες θέσεις, είναι πιο εργατικές, έχουν περισσότερες επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, παρόλα αυτά ε, υπάρχουν διακρίσεις στους μισθούς εις βάρος των γυναικών και μάλιστα οι εμπειρογνώμονες λένε ότι πολύ ακροθυγώς λαμβάνεται υπόψη στην οικονομική στρατηγική αυτή η διαφορά η μισθολογική. Αυτό ισχύει όχι μόνο για την Πολωνία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελειώνεται λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα εγκατακλείδη να πω ότι ένα επιπλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα η κυβέρνησή μας, είναι το θέμα της ε, μεταρρύθμισης, της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης και της εξίσωσης ε, του συνταξιοδοτικού ορίου ανδρών και γυναικών. Αναφέρεται ω κοινό ηλικιακό όριο για τη σύνταξη τα 67 χρόνια. Αλλά και αυτό είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλιά σας. Βέβαια, πιστεύω ότι αφορούσαν περισσότερο το δεύτερο πάνελ, το θέμα του δεύτερου πάνελ. Να σας υπενθυμίσω επίσης ε, ότι όσοι ευρωβουλευτές θέλουν το λόγο μπορούν να σηκώνουν το χέρι τους. Να σας παρακαλέσω και κάτι άλλο. Αν διαβάζετε με τέτοια ταχύτητα, ε, το ξέρω και από προσωπική πείρα, ότι ναι, μεν είναι εύκολο κανείς να διαβάζει με τρομερή ταχύτητα, αλλά για το διερμηνέ είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια. Δεν μπορεί να προλάβει. Γι' αυτό παρακαλώ να μιλάτε λίγο πιο αργά, για να μπορούν να σας μεταφράζουν. Ελιζαμπέτα Ράμπη, από την Ιταλική Γερουσία. Τρία λεπτά το πολύ. Και παρακαλώ τα θέμα, το θέμα σας ε, ουσιαστικά να αφορά αυτό του πρώτου πάνελ, αν είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για ένα θέμα σημαντικό. Σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική ημερίδα για τις γυναίκες ε, όλη τη οικουμένη. Στην Ιταλία, η συμμετοχή των ε, γυναικών στην αγορά εργασία σε καμία περίπτωση δεν έχει επιτύχει του στόχου τη ε, Λισαβόνα. Οι γυναίκε οι οποίε εργάζονται είναι 46,1%. Μιλάω για το 2010. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ βορρά και νότου της Ιταλίας. Διαπιστώνουμε ότι στο βορρά υπάρχουν πάνω από 56% ε, γυναική απασχόληση, αλλά στο Νότο το ποσοστό αυτό ούτε καν φτάνει το 30%. Οι γυναίκες εργάζονται κυρίως σε τομείς ε, με πολύ χαμηλές, ε, πολύ κακές αμοιβέ και αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με στερεότυπα του φύλου. Οι, τα δυνατότητες στα διδρομές είναι πολύ λίγες αλλά η θέση εργασίας σχετίζεται και με τις οικογενειακές υποχρεώσεις της γυναίκας στο πλαίσιο του νοικοκυριού. Παρά την καλή νομοθεσία, η πραγματικότητα, η καθημερινή πραγματικότητα λόγω της κρίσης βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις πολιτικές οι οποίες ε, εφαρμόζονται και για τη βελτίωση της γυναικείας απασχόλησης, αλλά και για τη συμφιλίωση, την πραγματική συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. οι γυναίκες και η οικονομία πλήτεται, πλήττονται λόγω του διαχωρισμού που παρατηρείται στην απασχόληση. Είναι ένας παράγοντας ανισότητας που επίσης ε, μειώνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος και τις δυνατότητε ανάπτυξης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι η Ιταλία στην Ευρώπη είναι η χώρα με τις περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες. Ο ορισμός ρόλων η διάκριση λόγω φύλου στην πρόσβαση εργασίας, στις συμβάσεις εργασίας, οι επιλογές επιμόρφωσης, εκπαίδευσης των γυναικών, ε, οι σταδιοδρομίες τους, ε, το πώς προχωρούν, πώς ανελίσσονται στην ε, ιεραρχία, την υπηρεσία... και θα πρέπει να σέβονται την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Όταν κάνουμε λόγο για στερεότυπα, για πολιτιστικούς, πολιτισμικούς παράγοντες, πρέπει να σας πω ότι ακόμη κυριαρχούν ε, στην κοινωνία μας, έχουν πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και αυτός ο οριζόντιος και κάθετος διαχωρισμός που υπάρχει στην αγορά εργασίας ουσιαστικά τιμωρεί τις γυναίκες αλλά και πτωχαίνει την κοινωνία που δεν μπορεί να αξιοποιήσει το μισό του δυναμικού ευφυΐας που διαθέτει οι συνθήκε εργασία των γυναικών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για την οικονομική ανάπτυξη και για τον ανταγωνισμό, αλλά και για να υπάρξει βελτίωση στην πολιτική ζωή, για να υπάρξει περισσότερη δημοκρατία στις χώρες μας. Εάν λοιπόν διεξάγουμε κάποιες εκστρατείες πληροφόρησης, πιστεύω ότι θα πετύχουμε την περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και τη μεγαλύτερη απασχόληση. Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, εάν γίνει, αλλά ακούγοντας και τις γυναίκες, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για τον εξυγχρονισμό της χώρας, για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων και για τις μελλοντικέ γένειες γυναικών. Στη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα σήμερα στην Ιταλία και η οποία αφορά τη μεταρρύθμιση των αγορών, Λέγεται ότι μία από τις μεγαλύτερες απαιτήσει είναι η βελτίωση των συνθήκων εργασίας για τις γυναίκες αλλά το ίδιο ισχύει για τις υπηρεσίες που προορίζονται για τις γυναίκες. Η Ιταλία, ολοκληρώνω, ολοκληρώνω, η Ιταλία έχει κάνει πολλά και στον τομέα των συντάξεων. Έχει γίνει σημαντική δουλειά για την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους. Θα πρέπει όμως να αποφύγουμε τη λήψη δρακόντιων μέτρων για να επιτύχουμε αυτή την ισότητα άνδρων και γυναικών. Πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία των γυναικών. Οι γυναίκες να μπορούν να επιλέγουν την ε, δουλειά τους με βάση τις ε, αρετές, τις ικανότητες, ε, τα προσόντα τους και να μπορούν έτσι να αναπτύξουν το όλο τους το δυναμικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω πλήρη κατανόηση ότι αυτός ο περιορισμός του χρόνου δεν είναι το ιδανικότερο. Το καταλαβαίνω, το ξέρω, αλλά παραδείγματος, παρακαλώ προσπαθήστε να μείνετε στα τρία αυτά λεπτά για να μπορούν όλοι να εκφράσουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους. Η κυρία Κρίστα Κλάους έχει το λόγο ευρωβουλευτές του σώματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για όσα ακούσαμε σήμερα το πρωί. Ακούσαμε πολλά καινούργια πράγματα και ήταν πολύ σημαντικό για μένα ε, το να ακούσω ότι άντρες ε, είναι σε καλύτερη θέση και χωρίς ε, δίπλωμα πανεπιστημίου από τις γυναίκες που έχουν το δίπλωμα. Δεύτερον, Άκουσα ότι έχουμε ένα διαχωρισμό των φύλων στην αγορά εργασία και αυτό δεν μου φάνηκε ότι ήταν θετικό. Και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία εκεί στο βήμα. Δεν το υποστηρίζουμε αυτό με όλες τις προσπάθειες που κάνουμε για κατανομή του προπολογισμού ανάλογα με το φίλο όταν ζητάμε στις γυναικών σε όλους τους τομείς. Δεν ξέρω, είναι φαύλος κύκλος. Πώς θα ξεφύγουμε. Και τρίτον, πώς αξιολογείται η, κατοίκον, η εργασία η οικιακή μάλλον. Υπάρχει μια ε, κοινωνική απόφαση που πρέπει να ληφθεί στην Ευρώπη, ελέγχθη. Αλλά αυτό είναι η κοινωνική απόφαση και των μεμονωμένων κρατών μελών. Και γι' αυτό εκπλήττομαι που ο Επίτροπος Λάσλο εκφράστηκε από αυτού. Αναφέρθηκε παραδείγματο χάρη όσον αφορά τα χρήματα για την ε, για τους παιδικούς σταθμούς στην Γερμανία. Γενικά έχω να πω ότι οι διάφορες δραστηριότητες στον κοινωνικό τομέα και στην, ε, η προσφορά υπηρεσιών στον οικιακό τομέα είναι το πιο, το πιο άνισο. Δηλαδή, εάν πληρώσει κανένας για την οικιακή εργασία είναι πανάκριβη. Αν την κάνει μόνος του δεν αξίζει τίποτα. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί μια καλύτερη αξιολόγηση της προσφοράς αυτής τη υπηρεσίας που προσφέρουν οι γυναίκες στην κοινωνία. Θα πρέπει κάτι να αξίζει και η εργασία αυτή και θα πρέπει για αυτό να φροντίσουμε και για τις γυναίκες που θέλουν να μείνουν σπίτι να είναι μητέρες, να είναι ε, στο περιβάλλον αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Χέλενα Διακό από την Ισπανική ε, Βουλή, ε, Γερουσία. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας συγχαρώ ε, για την θέση σας ε, ως Πρόεδρο της Επιτροπής. Ελπίζω να μην είναι εξαίρεση, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε και άνδρες ε, να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση για την ισότητα. Θα ήθελα να πω ότι στην Ισπανία τα τελευταία 30 χρόνια η αγορά εργασία στην Ισπανία έχει αλλάξει ριζικά και για ιστορικούς λόγους. Ενσωμάτωση, αγοράς ε, ε, στη, ε, γυναίκα στην αγορά, πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και το καθεξής. Αλλά βλέπουμε με τα στοιχεία ότι πολύ δρόμο έχουμε ακόμη να διανύσουμε. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Ισπανία Εξαιτία τη οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση επηρεάζει φυσικά του πιο ευάλωτου τομεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι ευάλωτη μόνο και μόνο επειδή είμαι γυναίκα. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η οικονομική κρίση και οποιαδήποτε εργασία και μεταρρύθμιση που μπορεί να ε, οδηγήσει απολύσεις ε, σε πιο αδύναμες μορφές συμβάσεων, φυσικά πλήττει άμεσα τους πιο ευάλωτους πολίτες. Γιατί οι γυναίκες δεν είναι κλάδος, είναι πολίτες. Ε, θα ήθελα να σας αναφέρω ένα στοιχείο που με ανησυχεί από ένα Ισπανικό Συνδικάτο, τη Γενική Ένωση Εργαζομένων. Αναφέρεται ότι με βάση τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι γυναίκες θα πρέπει να δουλεύουν 59 ε, μέρες περισσότερο από τους άνδρες για να κερδίζουν τις ίδιες ε, αποδοχές. Είναι μια χιονοστιβάδα, δηλαδή 59 μέρες περισσότερο θα πρέπει να δουλεύουν, που σημαίνει ότι κερδίζουν πολύ λιγότερο για την ίδια εργασία. Επίσης, είναι πολύ πιο εκτεθειμένες στην ανεργία ε, και είναι πολύ πιο εύκολο να μπουν οι γυναίκες στα γρανάζια για τι ανεργίε. Και στο μέλλον θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες για πρόσβαση σε σύνταξη, γιατί εξορισμού οι συντάξει των γυναικών είναι χαμηλότερε από τι συντάξει των ανδρών. Οπότε στην πρόταση ε, που μας έκανε μία από τις ε, εμπειρογνώμες του πάνελ, δηλαδή να καλέσουμε τους άνδρες ε, να μην πηγαίνουν στα πανεπιστήμια ή ή τις γυναίκες ε, να μην ε, σπουδάζουν ε, στα πανεπιστήμια. Είναι πραγματικά μια παράλογη πρόταση, αλλά πολύ σωστά το ανέφερε η προλαλή σας, γιατί θα μας βάλει σε σκέψεις. Αισθάνομαι υπερήφανη για τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν στην Ισπανία για θέματα ισότητας, για πάταξη της βίας μεταξύ των δύο φύλων και για τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας. Χαίρομαι για τις διατάξεις αυτές, αλλά ε, πολύ πρόοδο έχουμε ακόμη να σημειώσουμε και λυπούμε γιατί στην εποχή της κρίσης φαίνεται ότι οι γυναίκες θα είναι οι μεγάλες ξεχασμένες και στις διαδηλώσεις που γίνονται στην Ισπανία όλος ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Αν όμως το μοναδικό σύνθημα ε, της διαδήλωσης ήταν ε, για ίση και αξιοπρεπή απασχόληση για τις γυναίκες, δεν νομίζω ότι το, ο αριθμός των διαδηλωτών θα ήταν το ίδιο μεγάλος. Το λέω αυτό με απεσιοδοξία, αλλά και την αισιοδοξία ότι δεν είμαστε εμείς οι πιο ευάλωτες και ότι θα συνεχίσουμε με δυναμισμό τη μάχη μας. Ευχαριστώ. Το λόγο και ο κ. από την Βουλή της Ουγγαρίας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, χαιρετήσω ιδιαίτερα και εσάς, αλλά και τις γυναίκες συναδέλφους εδώ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη ε, τιμή που μπορώ να πάρω το λόγο σήμερα, όντας άντρας θα πρέπει να δούμε ε, τι γίνεται. Ε, στην ε, Βουλή στην Ουγγαρία έχουμε 9% μόνο γυναίκες και οι άντρες μέλη στη Βουλή γνωρίζουν τα προβλήματα αυτών των γυναικών και γενικά των γυναικών. Υπάρχει τώρα ένα νέο νόμος που λέει ότι οι γυναίκες είναι ισότιμες και προσπαθεί η Ουγγαρία να προωθήσει και να εγγυηθεί τα δικαιώματά τους, όπως και τα δικαιώματα ατόμων με δικές ανάγκες. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το γράμμα του νόμου θα γίνει πραγματικότητα μόνο εάν τα νομοθετικά όργανα περιέχουν μια ισότιμη εκπροσώπηση ε, ανδρών και γυναικών. Επίσης έχουμε την κάθετη και την οριζόντια ολοκληρώση. Υπάρχουν η, τα χαρακτηριστικά επαγγέλματα ανδρών, υπάρχουν οι, οι τυπικές θέσεις που μπορούν να πάρουν μόνο άντρες. Αλλά όταν ήδη στις βουλές της Ευρώπης οι αποφάσεις λαμβάνονται κυρίως από άντρες, πώς θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε αλλαγή. Η Γαλλίδα συνάδελφος Αγνής Παριτιών, στην οποία θα ήθελα να συγχαρώ, που είναι και μητέρα τεσσάρων παιδιών, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά συμφωνώ με αυτό που είπε ότι οι γυναίκες μετά από 8 ώρες εργασίας πρέπει να αναλάβουν ε, και άλλες εργασίες και είπε ότι θα χρειαστούν 40-50 χρόνια για να εξαλείψουν αυτές οι διαφορές. Είχε δίκιο ο συνάδελφος αυτό. Στην Ουγγρική Βουλή υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συζήτηση για την ισότητα και την ισοτιμία ανδρών και γυναικών. Και το μήνυμα του, της συζήτησης αυτής ήταν ότι χρειάζεται ριζοσπαστική αλλαγή και θα πρέπει να δούμε ποιο ήταν το όφελος της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτών των χωρών. Ο Πολωνός συνάδελφος είπε ότι προερχόμαστε από την ίδια περιοχή. Ναι, πραγματικά η κοινωνία ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και πολλές φορές οικονομικά δύσκολη και χάσαμε πολλά μετά την ένταξη. Στην Ουγγαρία με 7 εκατομμύρια κατοίκους χάσαμε 1 εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης μετά την ένταξη. Αυτό είναι το βάρος που έχουμε επομισθεί και δεν μπορούμε να πούμε ότι μας βοήθησε τόσο πολύ η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την θέση των γυναικών στην κοινωνία μας ε, με τέτοια προβλήματα στην αγορά απασχόλησης η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν οδήγησε σε επιτυχία στον τομέα αυτό και σε άλλους τομείς επίσης όχι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε πραγματικά ότι μειώθηκε η διαφορά ε, ανδρών και γυναικών στις παλιές αυτές ε, ε, στις νέες αυτές συγγνώμη χώρες του Ναντίον αυξήθηκε ιδίως επειδή αυξήθηκε και η ανταγωνιστική πίεση από τις χώρες της Δύσης. Είμαι, όπως σας είπα, περήφανος που στην Ουγγαρία οι διαφορές ε, των μισθών στην είναι μικρότερε μικρότερες από ό,τι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε και ο κ. Σούλτ, θα πρέπει να φροντίσουμε να εξαλειφθούν οι διαφορές αυτές. Και εκείνος αναφέρθηκε στην Γερμανία σε 20% διαφορά ενώ στην Ουγγαρία είναι μόνο 10%. Πολλές χώρες λοιπόν από την Ανατολική Ευρώπη έχουν προχωρήσει περισσότερο από ότι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικότερα έργα που πρέπει να επιτελεστούν πρέπει να εξαλειφθούν αυτές οι διαφορές. Ίσως υπάρχει κάποιος οδικός χάρτης, ίσως υπάρχουν εθνικές στρατηγικές, αλλά εφόσον οι, οι άντρες συμμαχούν μυστικά μεταξύ τους, δεν θα υπάρχει ποτέ καμία πραγματική πρόοδος. Πρό, πρόοδος. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που μιλήσατε και εσείς ε, ένας άντρας εδώ μεταξύ μας. Γιατί για μένα η ισότητα των φίλων δεν είναι θέμα των γυναικών. Όχι. Η ισότητα των φίλων είναι κάτι που αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αφορά δηλαδή και τους άντρες και τις γυναίκες που εξίσου πρέπει να μοιραστούν αυτή την ευθύνη να μοιραστούν τα δικαιώματα. Τώρα, έχω μια ερώτηση γιατί έχουμε τρεις ακόμα ομιλητές, αλλά δεν έχω τόσους πολλούς ομιλητές για το δεύτερο πάνελ η κυρία Αλίσσα Ολισόφσκα και η κυρία Πόπα Μικαέλα από την Πολωνία και από την Ρουμανία. Εσείς θέλετε να μιλήσετε για αυτό το πάνελ ή θέλετε να υποβάλλετε τι ερωτήσει στο επόμενο πάνελ. It's okay, next panel. Στο επόμενο, συμφωνείτε. Και οι δύο. Δεν βλέπω δύο απαντήσεις. Α, ωραία. Εντάξει. Ένας ομιλητής ακόμα. Από του εξωτερικού συμμετέχοντε. Η κυρία Ελίαν Χόφνερ από τη Σουηδία. Παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σήμερα οι γυναίκες έχουν πολύ καλή εκπαίδευση, παρόλα αυτά εξακολουθούν να παραμένουν οι άνδρες στις ε, υψηλότερες θέσεις και να κερδίζουν περισσότερα. Και πολλές φορές είναι δύσκολο οι γυναίκες να συμβιβάσουν τις διάφορες ε, υποχρεώσεις τους. Αναφερθήκατε στις μητέρες, δεν μπορεί κανένας να εργάζεται με πλήρη απασχόληση όταν τα παιδιά του είναι μικρά. Πολλές φορές οι γυναίκες εργάζονται με περιορισμένο χρόνο εργασίας, μερική απασχόληση δηλαδή, δεν μπορούν να κάνουν υπερορίες. Είναι αδύνατο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Δεν αρκεί δηλαδή να αναφερόμαστε μόνο στους μισθούς και να λέμε ότι θα πρέπει οι γυναίκες να ε, τύχουν σημείας μεταχείρισης. Ναι, αλλά στην πράξη τι γίνεται αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί και στον τόπο εργασία και στα σπίτια. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταία λέξη για την κυρία Στάινα Κάσακα από το, τη Βουλή της Λετωνίας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί συναδελφοί, δεν θα σηκωθώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Θα σας αναφέρω κάποια πράγματα για την Λετωνία. Σύμφωνα με την Ευρωστάτ, το 2002 στη Λετωνία οι γυναίκες ε, παίρναν 17,6% λιγότερο μισθό από ότι άντρες. Η διαφορά αυτή ε, είναι κατά 4,2 μεγαλύτερη από ό,τι ήταν δύο χρόνια νωρίτερα. Δηλαδή 17,6 το 2010. Το 2008 ήταν ε, διαφορετικό το επίπεδο αυτό. Περάσαμε το 2008 μια κρίση με διαφορετικές επιπτώσεις στην κοινωνία και η ανάκαμψη έγινε εις βάρος της κοινωνίας. Το Οικονομικό Φόρουμ προετοίμασε μια έκθεση για την κατάσταση στην Λετωνία και εκεί η Λετωνία βρίσκεται στην 19η θέση. Άμα δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες για εκπαίδευση, αλλά και η δυνατότητα της ε, πρόληψης στον υγειονομικό τομέα, βλέπουμε ότι για την πρόληψη στον τομέα της υγείας είμαστε οι πρώτοι Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Σε, ανάμεσα σε 135 χώρες η Λετωνία έχει τη θέση 22. Οι γυναίκες στην Λετωνία πρέπει να σας πω δεν εργάζονται τόσο πολύ σε επιχειρήσεις. Περίπου ο διπλάσιος αριθμός των διπλάσιος αριθμός ανδρών συγγνώμη, είναι επιχειρηματίες. Πριν από μερικά χρόνια αυτή η διαφορά ήταν ότι ήταν τριπλάσιο ο αριθμό των ανδρών. Έχουμε λοιπόν πετύχει κάποια πρόοδο. Το επόμενο πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι αυτή η αρχή της εισπληρωμής για την ίδια εργασία δεν είναι μεγάλο πρόβλημα στην Λετωνία γιατί όπως σας είπα οι γυναίκες εργάζονται κυρίως στον τομέα της προσφοράς υπηρεσιών ενώ οι άντρες ε, εργάζονται σε άλλους τομείς, επιχειρησιακούς τομείς. Και θα ήθελα για άλλη μια φορά να τονίσω ότι οι γυναίκες συνδέουν την επαγγελματική τους ζωή με άλλες υποχρεώσεις, παιδιά, παραδείγματο χάρη, τη φροντίδα της οικογένειας κλπ. Όσον αφορά τώρα το νομοθετικό πλαίσιο, έχω να πω ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την ε, ίση πληρωμή για την ίδια εργασία υπάρχει. Έχει διακανονιστεί το θέμα και πριν από ένα χρόνο εθετήθηκε και μια άλλη νομοθεσία, ένας άλλος νόμος που λέει ότι θα πρέπει το κράτος να ε, φροντίζει να υπάρχουν αρκετές θέσεις στα νηπιογωγεία για τα παιδιά από 1,5 ετών και πάνω. Τι συμβαίνει αυτό. Όσον αφορά τώρα την πολιτική ένταξη, έχω να πω ότι στην Βουλή της Λετωνίας υπάρχει 21% γυναικών. Στο Ευρωκοινοβούλιο 46%. Έχουμε λοιπόν αρκετή ε, οδό να διανύσουμε για να βελτιώσουμε την κατάστασή μας. Και τώρα ακόμα δύο λόγια για το πρόβλημα της ίσης πληρωμής για την ίδια εργασία. Υπάρχουν 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει μέσα η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να εξισώσει την κατάσταση και να πετύχει την ίδια ευημερία παντού. Και ίσως μία χώρα ε, παίρνει το ένα έβδομο της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι άλλες. Η χώρη μου, ιδίως όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές στην Γεωργία η Λετωνία παίρνει μόνο το 30% του μέσου όρου των πληρωμών της Ευρώπης στον τομέα αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ λίγο. Και βλέπουμε ότι οι γυναίκες δεν είναι τόσο ε, ευκίνητες, δεν έχουν την κινητικότητα που μπορούσαν να, να έχουν. Να θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε την ύπεθρο. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες παραμένουν φτωχές γιατί δεν έχουν τόσες δυνατότητες να εργαστούν. Αυτές οι άμεσες πληρωμές στη Γεωργία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικές για μας. το πρόγραμμα ε, μέχρι το 2020 ε, προβλέπει ότι θα αυξηθεί αυτό το ποσοστό από 30% στο 54% μόνο και εγώ θα ήθελα η ίση μισθή για η εργασία να ε, καλύπτουν όλους τους τομείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στο πάνελ θα δώσουμε το λόγο τώρα για τις τελευταίες παρατηρήσεις. Δεν ξέρω ποιος θέλει πρώτος να πάρει το λόγο. Yeah, reverse order maybe. Um, uh, uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Ε, κάποια σχόλια από πλευράς μου. Νομίζω ότι έχουμε κάνει δύο-τρεις πολιτικές επιλογές. Έχουμε αναλάβει κάποιες πολιτικές δεσμεύσεις, αλλά αυτές θα μεταφραστούν ε, σε πράξη μόνο αν αρχίσουμε να ε, συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα. Και για να το κάνουμε αυτό, πραγματικά πρέπει να υπάρχει και νομοθεσία, τα σχέδια στήριξης, Αυτά τα εργαλεία τα οποία αναπτύξαμε, όπως είναι η ενσωμάτωση της διάστησης του φύλου, πρέπει να μην είναι γραφειοκρατικά. Είναι σημαντικά εργαλεία που θα μας βοηθήσουν ε, να μετασχηματίσουμε την κοινωνία μας, να την κάνουμε όπως τη θέλουμε. Δεύτερο σχόλιο. Εάν θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης των γυναικών, πολλές από τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν θα βελτιώσουν ε, τις συνθήκες εργασίας για τους άνδρες και για τις γυναίκες από κοινού και κυρίως ε, θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των πιο ευάλωτων ατόμων. Πρέπει να πω ότι κάποια από τα εργαλεία που μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα δεν κοστίζουν δεν κοστίζουν, αλλά θα βελτιώσουν ε, την απασχόληση και την εργασία. Γιατί μιλάμε για βελτίωση του κοινωνικού κλίματο, μεγαλύτερη στήριξη, περισσότερη ηγεσία. Δεν κοστίζουν όλα αυτά. Και αυτά μπορούν να γίνουν ακόμη και εν καιρό κρίση. Είναι κάτι που θα βοηθήσει. Τρίτο σχόλιο, αυτό το παγκόσμιο ευρωπαϊκό μοντέλο. Πολλή συζήτηση έχει γίνει και με την Επιτροπή Στίγκλιτς για το πώς μετράτε το ΑΕΠΑ. Έχει γίνει συζήτηση για το κατά πόσον έχουμε τις σωστούς δείκτες που θα καθοδηγήσουν τις δράσεις μας. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη σχετική συζήτηση, το σχετικό προβληματισμό. Η μέτρηση της πρόνοιας είναι στο επίκεντρο, η ποιότητα ζωής, η ποιότητα εργασίας. Πρόκειται για σημαντικούς δείκτες. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι δείκτες είναι κατάλληλοι για να μπορέσουν να, να μας καθοδηγήσουν ε, στην εκπλήρωση των στόχων μας. Τέλος, η Ευρώπη νομίζω ότι Ήταν ε, σκαπανέας για την πρόθεση της ζήτηση για την ισότητα των φύλων. Έχει προωθήσει πολύ σημαντικά εργαλεία. Και σήμερα ακόμη περισσότερο είναι σημαντικό να συζητώνται τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις γυναίκες. Η Ανιέτα Στάρκ μίλησε για το τι παθαίνουν γυναίκες σε άλλες περιοχές του κόσμου. Έχουμε έναν ρόλο και ένα μοντέλο που πρέπει να το πρασπίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Το θέμα της ε, διάγνωσης και της γνώσης του τι συμβαίνει ενώ κάτι συμβαίνει είναι σημαντικό, πολλό δε μάλλον που αυτή η οικονομική αναδιάρθρωση λαμβάνει χώρα ραγδαία. Ακούσαμε πολλές παρατηρήσεις και σχόλια και για βελτιώσεις, αλλά και για επιδίνωση μετά την αναδιάρθρωση της οικονομίας. Είμαι πρόεδρος της ε, ε, Διεθνής Ένωσης για ε, φεμινιστές οικονομολόγους και έχουμε προγραμματίσει στη Βαρκελόνη την 21η καλοκαιρινή διάσκεψη τέλη του Ιουνίου. Εκεί θα εξετάσουμε θέματα της ε, συμπερίληψης της, ε, των ίσων ευκαιριών στον προπολογισμό, της ε, μισθολογικής διαφοράς, των συμβάντων στην Βόρεια Αφρική και στην Αγγής Ανατολή. Όλα αυτά θα τα εξετάσουν ε, γυναίκες οικονομολόγοι από τις ε, περιοχές αυτές. Επίσης, άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η διασύνδεση και ο συνειρμός ότι η αξία δεν αρκεί. Ε, και ε, η αξία <laughs> δεν είναι πάντα αρκετή, γιατί για να πληρώσει κανείς τις ανάγκες του χρειάζεται χρήματα. Δεν αρκεί να ασκεί ποιοτική εργασία. Και η διασύνδεση μεταξύ αξίας και αμοιβή είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα πρέπει να υπάρχει και ε, οικονομική αποτίμηση μιας αναγνωρισμένης αξίας συγκεκριμένη εργασία. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ δύσκολα, πολύ σύνθετα, αλλά πραγματικά κρίσιμα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έγινε και πολύ εύστοχες οι ερωτήσεις που ακούσαμε. Θα συνεχίσω από εκεί που τελείωσε η συνάδελφος. Το θέμα της αξίας και του χρήματος. Αξία και χρήμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Αυτό είπα και στην ομιλία μου, ότι 75% των ε, χαμηλότερων εισοδηματιών στην Ευρώπη είναι γυναίκες. Οπότε είναι τετάνιο το έργο που έχουμε να επιτελέσουμε. Θα ήθελα να σχολιάσω κάποια πράγματα. Ε, μ' αρέσουν ε, μερικά, μερικά συνθήματα που ακούμε και παραθέσεις. Ε, μερικές φορές όμως μου ακούγονται αστεία αυτά τα συνθήματα και τα τσιτάτα. Το, το πιο σημαντικό... Α, και, συγγνώμη, και το θέμα των ποσοστώσεων, οι ποσοστώσεις. Ε, οι ποσοστώσεις δεν είναι μόνο ε, στόχος, είναι και εργαλείο. Το θέμα είναι από τη στιγμή που υλοποιήσαμε το στόχο πρέπει να καταργήσουμε το εργαλείο. Όχι ακόμη θα έλεγα. Η ποσοστό είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και είναι πολύ εύκολο να ε, επανέλθουμε, να παραχωρήσουμε στην προηγούμενη αρνητική κατάσταση. Όπως είπε και η Ισπανίδα Συνάδελφο, είναι πολύ σημαντικό γιατί πραγματικά οι μεγάλε ξεχασμένε πολλέ φορέ στην κρίση είναι οι γυναίκε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι γυναίκε είναι τμήμα ε, της κρίσης και αντιμετωπίζουν στο πετσί τους πολύ έντονα αυτό το πρόβλημα. Βέβαια και οι άνδρες πλήττονται από την κρίση, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Θα ήθελα να σας πω κάτι που είπε ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, της πατρίδας μου. Είπε, δεν είναι ότι το πετρέλαιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για τον πλούτο της Νορβηγίας. Ε, οι γυναίκες είναι το πιο σημαντικό ο πιο σημαντικός πόρος, το πιο σημαντικό στοιχείο, γιατί ε, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόμενων στην ε, Νορβηγία, το 70% είναι γυναίκες. Βέβαια, πολλές εργάζονται σε μερική απασχόληση, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε υλοποιήσει το στόχο της πλήρους απασχόλησης. Πάντως, όταν έχουμε ένα καλό σύστημα πρόνοιας, όταν επενδύουμε στις γυναίκες, ε, επενδύουμε ουσιαστικά στην ε, κοινωνική μας ανάπτυξη. Δεν νομίζω να είναι εκλειφθεί ως αλαζονικό, από ότι το σκανδιναβικό μοντέλο πρόνοιας είχε και ένα άλλο αποτέλεσμα. Έχει και πολύ ψηλό ποσοστό ε, γεννητικότητας και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ και τις τρεις ομιλητρίες του πάνελ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και συνεισφέρατε στην σημερινή μας ε, συζήτηση. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο πάνελ. Ευχαριστώ και πάλι. Uh, στο δεύτερο τμήμα της ημερίδας θα συζητήσουμε τρόπους ε, για να συρρυκνωθεί το χάσμα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Θα ανταλλάξουμε εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και αφού ακούσουμε καταρχάς ε, έναν γύρο ομιλιών, θα μπορέσουμε να ακούσουμε εθνικές ε, εμπειρίες και πρακτικές. Να μην χάνουμε χρόνο λοιπόν. Να δώσω στο, το λόγο καταρχάς στην κυρία Αλένα Γκαϊντούσκοβα, αντιπρόεδρο της Γερουσίας στην Τσεχική Δημοκρατία. Πέντε λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την διοργάνωση της σημερινής συνεδρίασης. Ένα θέμα άκρος επίκαιρο σήμερα στην Τσεχία. Αποτελεί τιμή για μένα απλαμβάνω λαμβάνω το λόγο εδώ, αν και η κατάσταση στη Τσεχία συχνά είναι ένα αρνητικό παράδειγμα σε ό,τι αφορά τις μισθολογικές διαφορές. Η χώρα μας έχει μία από τις μεγαλύτερες ε, μισθολογικές διαφορές μεταξύ άνδρων και γυναικών ε, που αγγίζει το 26%. 8 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω, αντιδρώντας ε, και σε αυτά που είπε πριν από εμένα πρόσωπο της Ουγγαρίας, αυτές οι διαφορές ε, σημαντικά αυξήθηκαν ε, με τις δεξιές κυβερνήσει και όχι μετά την προσχώρηση της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα έγινε αυτό και ήταν συνέπεια της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και ιδεολογίας φαίνεται να είναι ε, δικαίωμα του εργαζομένου στη χειρότερη περίπτωση και ηθικά αποδεκτό στην καλύτερη το να υπάρχει διάκριση ε, τέτοιου είδους κατά των γυναικών. Υπάρχουν ε, Επίσης, πολλές περικοπές σε αυτή την περίοδο στις θέσεις μερικής απασχόλησης, στις αργασιακές σχέσεις, βλέπουμε μεγάλη επιδείνωση και όλα αυτά εμβαθύνουν το χάσμα στις αμοιβέ ε, των γυναικών σε σχέση με τις αμοιβέ των ανδρών. Σήμερα γίνεται μεγάλος λόγος στα μέσα ενημέρωσης ε, για τις ε, διαφορές της αμοιβέ, αλλά κυρίως οι ακαδημαϊκοί και μη κυβερνητικέ οργανώσεις συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Όχι η πολιτική, όχι η κοινή γνώμη. Νομίζω ότι μόνο με οικονομικά επιχειρήματα ε, θεωρούν οι νοφιλεύθεροι ότι μπορούμε να πετύχουμε. οικονομική πτυχή, η οικονομική συνιστόσα μπορεί μόνο να πετύχει αλλαγή. Εγώ θέλω να προτείνω μια διαφορετική γραμμή επιχειρηματολογίας. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός ε, περιβάλλοντος εργασιακού που δεν ε, συνιστά διακριτική μεταχείριση. Αν δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση, μπορούν οι επιχειρήσει ε, να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά και να αποκτήσουν το πλέον ε, προσοντούχο εργατικό δυναμικό. Σε πολλέ έρευνε σήμερα βλέπουμε ότι οι εταιρείε ε, προωθούν τις ίσες ευκαιρίες, άρα έχουν άτομα με περισσότερα κίνητρα ως υπαλλήλου, με μεγαλύτερη ικανοποίηση και παραγωγικότητα. Άρα βελτιώνεται και η εμπορική εικόνα τους, το εμπορικό τους σήμα. Επίσης θα ήθελα να πω για τα πλεονεκτήματα που έχει η κατάργηση των διακρίσεων στην εργασία γενικότερα για την κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο εθίγει και στην προηγούμενη συζήτηση. Η άρση του χάσματος της αμοιβέ θα βελτιώσει και την κατανάλωση αλλά και την παραγωγικότητα στην κοινωνία και έτσι θα λυθούν τα προβλήματα της διαρθρωτικής ανεργίας των γυναικών και όσο είναι στην παραγωγική ηλικία και αφού συνταξιοδοτηθούν. Επίσης, αν υπάρχει μεγαλύτερη εισφορά λόγω και του εισοδήματο των γυναικών, αυτό βελτιώνει το σύστημα υγείας και τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρικοδοτούνται. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό νέο, αλλά οι πρωταγωνιστές ε, στην Τσεχία έχουν διαπιστώσει ότι ίσες ευκαιρίες δεν είναι μόνο τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή κάποια κοινωνικά προγράμματα, αλλά ότι υπάρχει και το στοιχείο της επιχείρησης. Ίσως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το αρνητικό πολιτικό κλίμα και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όταν μιλάμε για χάσμα στις αμοιβέ ανδρών και γυναικών, να μην ξεχνάμε και άλλες δύο μορφές διάκρισης ε, των γυναικών στην αγορά εργασίας. Πρώτα απ' όλα, συμφιλίωση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Δεύτερον, ε, στερεότυπα για το ρόλο ανδρών και γυναικών στην κοινωνία. Διαστάσεις αλληλένδετες μεταξύ τους. Έχουν αναφερθεί στην προηγούμενη συζήτηση αυτά τα θέματα. Άρα, αν θέλουμε να συρρυκνώσουμε το χάσμα στις αμοιβέ, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και τις δύο άλλες μορφές διάκρισης που σας προανέφερα. Στην Τσεχική Δημοκρατία έχουμε τον νόμο κατά των διακρίσεων, σύμφωνα και με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική, όπως προείπα. Αυτό που θέλω πάντως να πω είναι ότι η νέα γενιά των πολιτικών μας είναι αυτοί που όπως πάντοτε τους λέω θα πρέπει να θέσουν κανόνες που θα άρουν τις διακρίσεις κατά των γυναικών. Ακόμη και στη ζυγική δημοκρατία που βελτιώνεται η κατάσταση των γυναικών που καταφέρουν οι γυναίκες να καταλάβουν αξιώματα με υψηλότερη αμοιβή πάλι πιστεύω ότι θα πρέπει να ισχύουν ε, οι, οι νόμοι. Βέβαια δεν θα πρέπει να φτάσουμε και στο άλλο άκρο με τους νόμους κατά των ε, διακρίσεων. Για να πετύχουμε την αηφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας πρέπει να κινητοποιήσουμε ολόκληρο το δυναμικό της κοινωνίας. Το παράδειγμα της Νορβηγίας είναι πάρα πολύ καλό. Όταν έχουν όλοι και όλες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους ε, σε πνεύμα συνεργασίας και σε αρμονικές σχέσεις. Έτσι θα έπρεπε να τα πράγματα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα να συνεισφέρω και εγώ στην αποψινή, στη σημερινή μάλλον συνεδρίαση. Να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου στην προσπάθεια για μεγαλύτερη, για πραγματική ισότητα. Να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο, ιδίως τον πρόεδρό του, τον Μάρτιν Σούλτ, που είναι η αιχμή του δόρατο αυτής της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία. Thank you very much for that. Ευχαριστώ. Παίρναμε τώρα στην επόμενη ομιλητριά μας, την κυρία Ντορίνα Μπιάνκη, που είναι μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης ε, της Τελικής Γερουσίας. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη αυτή ευκαιρία που δίνεται στην Ιταλική Βουλή και συγκεκριμένα στην Ιταλική Γερουσία να συμμετέχει στον πολιτικό διάλογο με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα στα πλαίσια της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Επιτροπής, όχι μόνο ως πρόεδρο αλλά και ως άνδρα, γιατί είμαι πεισμένη ότι ε, είναι σημαντικό να συμμετέχουν ε, οι άνδρες σε αυτή τη συζήτηση. Είναι σημαντική η συμμετοχή τους, ε, έχει αποφασιστική σημασία για την βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Όπως σημαίνει και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ιταλία, παρά την κατάλληλη εθνική νομοθεσία, διαπιστώνουμε μία μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών σημαντική. Και μάλιστα το μισθολογικό χάσμα στην Ιταλία είναι αντίστοιχο με άλλων χωρών. Ε, παρόλο που έχουμε ίδια εργασία, οι άντρες κερδίζουν περισσότερο. Ε, και δυστυχώς οι γυναίκες αμείβονται με χαμηλότερους μισθούς, παρόλο που επιτελούν παρόμοια εργασία. Ε, οι λόγοι είναι πολύ και διάφοροι. Έχουμε διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, όπως είπαμε προηγουμένως. Ε, ακόμη και σήμερα άνδρες και γυναίκες έχουν διαφορετικά επαγγέλματα και κάνουν διαφορετικές εργασίες και οι γυναικείες εργασίες υποβαθμίζονται. Επίσης οι μορφωτικές διαφορές ε, επηρεάζουν το προφίλ και τη σταδιοδρομία. Ε, το θέμα του συνδυασμού της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Επίσης το θέμα των φροντίδων και οικογενειακές υποχρεώσεις που δεν κατανέμονται κρυβοδίκαια μεταξύ ανδρών και γυναικών όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα και, στο, ε, και στην γονιμότητα και στην υπογεννητικότητα. Ε, σίγουρα η παρουσία παιδιών επηρεάζει αρνητικά την ε, μισθολογική εξέλιξη των γυναικών. Αναφέρεται από την Εθνική Υπηρεσία ότι δυστυχώς η Ιταλία πόρα απέχει από την τήρηση των ε, ευρωπαϊκών στόχων για την ίση απασχόληση ανδρών και γυναικών. Σίγουρα η γυναική ανεργία είναι πολύ ψηλότερη από την ανδρική. Επίση, οι γυναίκε προσφεύγουν πολύ περισσότερο στην μερική απασχόληση, όπω μα είπαν και οι προλαλήσαντε. Έχουμε περισσότερε ε, ε, γυναίκε στι ατυπικέ μορφέ εργασία. και δυσκολεύονται οι γυναίκε να συμφιλειώσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Έτσι, Ιδιαίτερα όταν έχουμε μικρά παιδιά, οι γυναίκες απασχολούνται όλο και λιγότερο. Οι γυναίκες, ε, όπως είπαμε, έχουν ε, πολύ πιο χαμηλά εισοδήματα και εκπροσωπούνται πολύ λιγότερο σε υψηλά κλιμάκια ή διευθυντικές ε, θέσεις. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σε ορισμένες χώρες. Επίσης, η, η χαμηλότερη αμοιβή των γυναικών έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Παρά τις ε, επιδοτήσεις που δίνονται και ορισμένα οικογενειακά επιδόματα. Αυτά, φαίνονται, αυτά όλα φαίνονται και σε κάποια στοιχεία για τις μισθολογικές διαφορές ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών για το 2010. Πρόκειται για στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι στην Ευρώπη, στις 27 χώρες μέλη, ο μικτός ε, μισθός των γυναικών ήταν κατά 16,4% χαμηλότερος από το μεικτό ανδρικό μισθό. Στην ε, Ιταλία Η διαφορά είναι 5,5% σε αντίθεση με το 15% ε, στην Σουηδία ή το 4% στη Φιλανδία. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάσταση είναι καλύτερη στην Ιταλία. Απλώς ε, ε, δουλεύουν πολύ περισσότερες γυναίκες στην Ιταλική αγορά εργασίας από ό,τι σε άλλες χώρες και επίσης έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό γυναικείας ανεργίας, ιδιαίτερα στις ανειδίκευτες θέσεις. Παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις στην Ιταλία που είναι πολύ σύγχρονες, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί αισθητά. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλές νομοθετικές διατάξεις υπέρ της ίσης μεταχείρισης των γυναικών και ε, ίσης αμοιβής. και μάλιστα τα τελευταία παρέμβαση ήταν το διάταγμα της ε, Επιτροπής Απασχόλησης του 2010 για ε, ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ε, παρότριση προς την ε, Ιταλική κυβέρνηση να εφαρμόσει και εμπράκτο στο σχέδιο δράσης ε, Ιταλία 2020 και να, να εφαρμοστούν εμπράκτος οι ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Η Οδηγία 54-2006 ενσωματώθηκε στην Ιταλική Ένωμη Τάξη με ένα νομοθετικό διάταγμα όπου προσδιορίζονται κάποια άρθρα του κώδικα ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και εκεί προσδιορίζεται η άμεση και άμεση διάκριση στο χώρο εργασία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μισθολογική διάκριση, είτε άμεση είτε έμεση, για ίδια ή εισάξια εργασία. Και επίσης ε, απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλους, οποιαδήποτε άλλους διάκριση στον εργασιακό χώρο. Επιβάλλονται μάλιστα ε, κυρώσει σε περίπτωση που παραβιάζονται αυτές ε, οι διατάξεις κατά των διακρίσεων. Και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ε, μπορεί να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την πάταξη των διακρίσεων και προβλέπεται ο διορισμός συμβούλου ισότητας ευκαιριών σε εθνικό, περιφερειακό και επαρχιακό επίπεδο. Σήμερα στην Ιταλία τα συνδικάτα και η Ιταλική Βουλή ασχολούνται με το θέμα της εργασιακής μεταρρύθμισης. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις τη μισθολογική κατάσταση των γυναικών. Αυτό είναι σημαντική διεκδίκηση της Ιταλικής κοινωνίας. Να μην ξεχάσω και το χάρτη ισότητας ευκαιριών και ισότητας στο χώρο εργασίας που κυρώθηκε τον Νοέμβριο του 2009 στην Ιταλία και μάλιστα έχει ε, υπογραφεί από πολλές εταιρείες και επιχειρήσεις. Παρακαλώ ολοκληρώστε γιατί έχετε εξαντλήσει το δίλεπτο που δικαιώσασταν. Α, νομίζω ότι είχα περισσότερο χρόνο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ήταν πέντε λεπτά ο χρόνος σας. Αλλά έχετε κατά δύο λεπτά τον έχετε ξεπεράσει κατά δύο λεπτά. Θα ήθελα να μιλήσω για ένα νέο νομοσχέδιο που συζητάτε το τελευταίο χρόνο στην Ιταλία και αφορά τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις Μάλιστα εκεί προβλέπετε ότι οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείε έχουν υποχρέωση να απασχολούν μέχρι το 2015 30% και 40% ε, μέχρι το 2014 γυναίκες, να απασχολούν γυναίκες. Νομίζω ότι αυτή η νομοθετική διάταξη, αυτός ο νόμος είναι πολύ σημαντικός και μάλιστα έχει ε, περάσει και από τη Βουλή και από τη Γερουσία και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αλλαγή στην ε, Ιταλική νομοθεσία. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω μια φράση που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε από το καταπληκτικό μυθιστόρημα της ε, Virginia Woolf ότι σήμερα δηλαδή ε, η σημασία της οικονομικής ανεξαρτησίας και αυτονομίας ε, των γυναικών είναι πολύ σημαντική. Αυτό το επισήμανε και οι προλαλήσαντες και τα μέλη του πάνελ και νομίζω ότι από αυτό εξαρτάται και η μελλοντική εξέλιξη της κοινωνίας μας. Θα πρέπει ο ρόλος των γυναικών να αναδειχθεί δεόντως για να πετύχουμε μια πραγματική ισότητα των δύο φύλων. Αυτό μας ενδιαφέρει, μια οικονομική ανεξαρτησία, αλλά και μια σωστή μελλοντική οργάνωση των κοινωνιών μας. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στον επόμενο ομιλητή. Η κυρία Τέρα Αλγουρία, μέλος της Επιτροπής ε, ε, Θεσμικών Θεμάτων της ε, Πορτογαλικής Βουλής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Καταρχήν είναι τιμή μου και ευχαρίστηση που είμαι εδώ. Ελπίζω ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Η κοινωνική διάσταση της ανισότητας είναι όσο πάει και πιο εμφανής. Από την προοπτική του, του φύλου, η ισότητα ανδρών και γυναικών σημαίνει τροποποίηση των κοινωνικών ρόλων ανδρών και γυναικών. Ο στόχο βέβαια δεν είναι να ανηθούμε τι διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ των φύλων, αλλά να εξαλείψουμε τι ασυμμετρίε που οφείλονται σε κάποιους κοινωνικούς ρόλους. Το πιο ενδιαφέρον είναι ακριβώς αυτό. Να καταλάβουμε ότι έχουμε κάποιες κοινωνικές σχέσεις που βασίζονται στα φύλλα που είναι ασταθείς και εξακολουθούν να επανορίζονται κάθε φορά χωρίς να είναι κάτι που είναι πραγματικά οριστικό και σταθερό και βασίζεται κυριολεκτικά στο, στη φύση. Θα πρέπει να υπάρχει ίση αμοιβή για ίση εργασία. Οι διαφορές οι μισθολογικές μεταξύ ανδρών και γενικών είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας ανισότητας. Ε, θα έπρεπε άντρες και γυναίκες ε, να δούμε ότι όχι μόνο πληρώνονται διαφορετικά εις βάρος των γυναικών για την ίδια εργασία, αλλά ταυτόχρονα απασχολούν σε διαφορετικές ε, απασχολώσεις που εργασίες που χαρακτηριστικά γίνονται από γυναίκες πληρώνονται γενικά χαμηλότερα από εκείνες που γίνονται συνήθως από άντρες. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι μια βασική αρχή του Πορτογαλικού Συντάγματος και ένα από τα κύρια έργα της, του κράτους είναι να την εφαρμόσει αποτελεσματικά με την οθέτηση των σχετικών δημοσίων πολιτικών. Η εξάλληψη κάθε μορφής ε, διακρίσεων κατά των γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντική για την ποιότητα της δημοκρατίας και την ανάπτυξη. Και νομικά και ε, συνταγματικά η θέση των γυναικών είναι ιδιάζουσα. Ο πρόεδρος διακόπτη πρέπει να μιλάτε λίγο πιο αργά παρακαλώ, Αλλιώ δεν μπορούν να σα παρακολουθούν οι διερμηνείς. Μάλιστα. Λοιπόν, το ποσοστό τη απασχόληση γυναικών, παραδείγματο χάρη, είναι ιδιαίτερα υψηλό στην Πορτογαλία. Οι περισσότεροι φοιτητέ και οι πιο επιτυχεί ε, στα πανεπιστήμια είναι οι γυναίκε. Ε, επιστημονικές και τεχνικές εργασίες επίσης κατέχονται από γυναίκες. Παρ' όλα αυτά όμως άλλα κοινωνικά στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα της χώρας. Οι μισθοί είναι συνήθως χαμηλότερες, οι οικιακές εργασίες δεν κατανέμονται και γίνονται κυρίως από τις γυναίκες και ο δημόσιος τομέας ε, βρίσκεται κάτω την ε, επίδραση των κομμάτων στο οποία λείπουν οι γυναίκες. Δηλαδή υπάρχει μία α, αντίφαση ανάμεσα στους νόμους και στην πράξη στην Πορτογαλία. Το συνταγματικό και νομικό σύστημα έχει σαν στόχο κάποιο διακανονισμό που ε, δίνει στις γυναίκες τη πραγματική του αξία. Παρ' όλα αυτά, ταυτόχρονα υπάρχει μια κοινωνική πτυχή που συνήθως οι γυναίκες την αποδέχονται και που είναι εις βάρος τους είναι αντίθετη με το ε, ιδανικό της χειραφέτησης. Και αυτό μπορεί να το δείτε στην ε, αδυναμία των ανεξαρτήτων ε, κοινωνικών κινημάτων που έχουν σαν στόχο μία αλλαγή εκ των άνω προς τα κάτω του του βέβαια θα πρέπει να δούμε πώς η επιβολή παρεμποδίζεται από τις ιδέες της διάκρισης στη κοινωνία γενικά. Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα στην Πορτογαλία είναι ακριβώ η διαφορά μεταξύ της νομοθεσίας και του συντάγματος αφενός και της ε, καθημερινής πραγματικότητας αφετέρου. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερο στη συγκέντρωση την υψηλή των γυναικών σε λίγες μορφές, σε λίγα επαγγέλματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας ενδυναμώνοντας και προσαρμόντας τις απαραίτητα σώματα ισότητας που υπάρχουν. Ο πρώτος διακόπτη πάλι μιλάτε πάλι ξανά πολύ αργά. Ε, γρήγορα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε την αγκαιότητα συλλογή στοιχείων. Οι περισσότερε έρευνε θα πρέπει να γίνουν με πάντα τον παράγοντα του φύλου. Θα πρέπει επίση να ενθαρρυνθεί περισσότερη έντονη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των διαφόρων οργανώσεων για την πρόσπιση των δικαιωμάτων αυτών. Το πρόγραμμα του 19ης Συνταγματικής Κυβέρνησης τονίζει πόσο σημαντικό είναι η επίτευξη και προώθηση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων στην κοινωνία, τονίζοντας την ισότητα ανδρών και γυναικών όχι μόνο σαν θέμα δικαιωμάτων και κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και σε μια προϋπόθεση για την επίτευξη αηφόρου ανάπτυξης, απασχόλησης και αλληλεγγύης. Υπάρχουν πλεονεκτήματα αν υπάρχει ισότητα στην νομοθεσία και υπάρχουν πολλά βήματα που αναλαμβάνουν για να επιτευχθεί η ισότητα αυτή. Στην ε, Πορτογαλία όσον αφορά την πολιτική συμμετοχή άνθρωπων και γυναικών έχουμε τη μεγαλύτερη ισότητα. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο όμως για την εκπροσώπηση και των δύο φύλων στη ε, λήψη οικονομικών αποφάσεων όπου η παρουσία των γυναικών είναι επαρκή. Για να αλλάξει η κατάσταση αυτή, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας την περασμένη εβδομάδα υιοθέτησε ένα ψήφισμα που απαιτεί από εταιρείε του δημοσίου τομέα να εγκρίνουν ε, διατάξεις για την ισότητα, ούτως ώστε να πετύχουν την ισότητα ανδρών και γυναικών στις επιχειρήσεις. Το ίδιο θα ζητηθεί επίσης και για ιδιωτικές επιχειρήσεις και η εξολόγηση γίνεται από το κάθε έξι μήνες. Η Πορτογαλική Βουλή είχε σημαντικό ρόλο να παίξει όσον αφορά την εποπτεία αυτών των νόμων, ιδίω μέσω τη Υποεπιτροπή για την Ισότητα. Ταυτόχρονα όμω θα πρέπει να προωθήσει τη συζήτηση και να συμβάλλει στην ε, αφύπνιση τη κοινωνία. Το έκανε στο παρελθόν και θα το κάνει και στο μέλλον. Τέλο, θα ήθελα να αναφερθώ στι δύσκολε στιγμέ ε, που ζούμε αυτή τη στιγμή και τι επιπτώσει για τι γυναίκε. Στη βαθιά αυτή η οικονομική κρίση που ήδη αναφέρθηκε. Έχουμε βέβαια πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην πρόοδο της ισότητας γιατί η απασχόληση σε ε, ευάλωτες θέσεις ε, ε, απασχόλησης εκθέτουν τις γυναίκες περισσότερο στην κρίση αυτή. Δηλαδή, με δύο λόγια, πολλά έγιναν, πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν. Οι βουλευτές έχουν πολύ σημαντική ευθύνη. Το έργο του δεν ήταν δύσκολο ούτε στο παρελθόν, ούτε είναι σήμερα, ούτε θα είναι στο μέλλον. Τούτων εχθένων σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank uh, Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε παρουσιάσεις από εκπροσώπους τριών διαφορετικών κοινοβουλίων. Και περνάμε τώρα στον κατάλογο των ομιλητών. Να πω όμως πρώτα ότι περιμένουμε την Επίτροπο Ρέντινγκ. Έχει μόνο μισή ώρα στη διάθεσή της να μας αφιερώσει. Άρα όλοι τα ανέρθα ως αμέσως το λόγο. Μέχρι να έρθει όμως να δώσω το λόγο στην κυρία Λύσια Ολυσόσκα από την Πολωνική Βουλή. Σας παρακαλώ όμως να είστε σύντομοι, γιατί έρχεται όπου να είναι και η κυρία Ρέντινγκ. Παρακαλώ, σας δίνω το λόγο, έχετε τρία λεπτά. ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μία γυναίκα που έχει επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα, πολύ ευχαρίστως βοηθά ε, και στην τοπική αυτοδιοίκηση, και στα... θέλει να συμμετέχει στην κατάρτιση νέων μαθητευόμενων που ψάχνουν δουλειά μέσω των γραφείων απασχόλησης. Είναι πολύ αφοσιωμένη και αξιολογεί και ενισχύει τις νέες γυναίκες που ψάχνουν δουλειά. Βέβαια υπάρχουν διαφορές ε, ε, από τις ε, γυναίκες που είναι διευθυντήρες. Από το, οι γυναίκες διαφέρουν από τους άντρες όταν έχουν ε, διευθυντικές θέσεις. Γιατί οι άντρες δεν ε, συμπεριφέρονται αντίστοιχα προσπαθώντας να βοηθήσουν τους υπόλοιπους άντρες. 54%, 54 των γυναικών απασχολούνται στην Πολωνία, αλλά δυστυχώς η συμμετοχή στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ χαμηλότερη και δυστυχώς δεν τηρούνται οι ε, διατάξεις του εργατικού κώδικα. Είναι πολύ ε, εύκολο να ε, διαπιστώσει μια γυναίκα που επιστρέφει από άδεια μητρότητα ότι υποβαθμίζεται η θέση απασχόλησης, της, την μεταθέτουν σε χαμηλότερες ε, θέσεις. Επίσης, ακόμη και αν κρατάει λίγο η άδεια μητρότητα για τη γυναίκα, είναι πολύ δύσκολο να μην διαπιστωθεί επιδείνωση στους, όρους, ε, στους εργασιακούς της όρους. Έχουμε δυσάριστη κατάσταση στις γυναίκες ό,τι αφορά και την ε, λήψη δανείων για γυναίκες που μόνες τους ανατρέφουν ε, τα παιδιά τους, που μεγαλούν τα παιδιά τους, είτε είναι ένα είτε περισσότεροι. Υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα, αλλά όχι μόνο οικονομικά προβλήματα για τις γυναίκες. Και από ηθική άποψη αισθάνονται ε, υποβαθμισμένες οι γυναίκες γιατί ε, δεν έχουν ίσες δυνατότητες λήψης δανείων. Τι μηχανισμούς λοιπόν θα πρέπει να υιοθετήσουμε στις γυναίκες αυτές που δυστυχώς ε, είναι μόνες τους και μόνες τους είναι υποχρεωμένες να θρέψουν τα παιδιά τους να έχουν ίσες συνθήκες πρόσβασης στην καταναλωτική πίστη και στα δάνεια γιατί είναι μια επιπλέον ε, δυσκολία αυτή για τις γυναίκες, η οικονομική δυσκολία. Οι, γυναί... οι άντρες πολύ πιο εύκολα έχουν πρόσβαση στο δανεισμό, οπότε η χειραφέτηση γίνεται στην πράξη πολύ πιο δύσκολη. Το οικονομικό θέμα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και ε, είναι πολύ δύσκολο για τις γυναίκες μόνες τους να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα όταν μόνες τους αναθρέφουν τα παιδιά τους. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ. Thank you very much. And, uh, the floor Ευχαριστώ πολύ κυρία Πόπα Χαίλκα από την Γερουσία της Ρουμανίας. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να ε, ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά για την ε, σημερινή γιορτή της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας και να πω ότι στα θέματα ισότητας δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ποσότητα αλλά και η νομιμότητα. Η παιδεία, η εκπαίδευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξει η νοοτροπία. Εγώ σπούδασα μαθηματικά και όταν σπούδαζα ήμασταν στο μαθηματικό τμήμα μόνο τρεις γυναίκες. Σήμερα 40% των γυναικών στρέφονται προς ε, τεχνικούς τομείς που σπουδάζουν στις θετικές επιστήμες. Φαίνεται ότι έστω και αργά η νοοτροπία αλλάζει. Βέβαια, δυστυχώς ε, υπάρχει μισθολογικό χάσμα και διευθυντικές θέσεις ε, δεσπόζονται κυρίως από άνδρες. Και υπάρχουν και επαγγέλματα που είναι κατά παράδοση ανδροκρατούμενα, η πολιτική για παράδειγμα. Θα μπορούσα να σας δώσω ένα παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στη Ρουμανία. Η πρόεδρος της Βουλής είναι γυναίκα. Ε, η Γενική Εισαγγελέα ε, στην ε, Ρουμανία είναι γυναίκα επίσης. Και μάλιστα ως πρώην Ευρωβουλευτής θα περίμενα και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να γίνει γυναίκα. Υπάρχει δυστυχώς μεγάλη απόσταση πολλές φορές μεταξύ θεωρίας και πράξης. Χρειαζόμαστε κάποιες κοινοτικές πολιτικές ε, είναι πολύ πιο σημαντικές οι πανευρωπαϊκές πολιτικές από τις εθνικές πολιτικές για τη συρρήγνωση αυτού του μισθοδολογικού χάσματος. Επαναλαμβάνω, ε, ετοιμάζουμε και καταρτίζουμε νέους για να εργαστούν στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο προσόντων και δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Γιατί λοιπόν να μην ε, προταθούν και ε, νέα μέτρα στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ας σκεφτούμε τους νέους, ας ενθαρρύνουμε μια μεταστροφή της νοοτροπίας. Πολλές φορές έχουμε φαινόμενα σώματεμπορίας και ε, εργασίας σε πολύ υποβαθμισμένες συνθήκες, ουσιαστικά σε συνθήκες ε, υλωτίας. Θα πρέπει τέτοιες πρακτικές να παταχθούν. Στη Ρουμανία η μισθολογική διαφορά ευτυχώς έχει μειωθεί από 21% το 1994 σε 12% το 2009. Και έχουμε και μερικές περιπτώσεις ε, καλών πρακτικών. Η Ρουμανική Γερουσία, για παράδειγμα, διοργάνωσε μια ε, εθνική ημέρα ίσης ε, αμοιβής ανδρών και γυναικών και η Επιτροπή Ισότητας Ευκαιριών πρωτοστάτησε στην διεξαγωγή μιας ε, εκστρατείας για τις γυναίκες στην Ήπεθρο και για την εθάρρηση του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ήπεθρο. Έχουμε μάλιστα και έναν εθνικό φορέα για την ισότητα των ευκαιριών. Ε, ο φορέας αυτός ε, προσπαθεί να συμβάλλει σε μια αλλαγή της νοοτροπίας, ε, να δώσει κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για τις πολιτικές και να φέρει τις γυναίκες στην πολιτική, βελτιώνοντας επίσης τη θέση των γυναικών και στην Ήπεθρο. Στην Ρουμανία έχουμε μόνο 7 γερουσιάστριες, 6% δηλαδή της ε, ρωμανικής γερουσίας. Οπότε φαίνεται ότι η ρουμανική κοινωνία δεν είναι ακόμη έτοιμη έτοιμη να ψηφίσει γυναίκες. Εφαρμόζεται το σύστημα του Σταυρού. Επαναλαμβάνω, η πολιτική είναι ένας από τους κλάδους που είναι καταξοχήν ανδροκρατούμενοι. Διαρωτώ με λοιπόν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει ε, προτάσεις για την αποκατάσταση της ισότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κατέθεσε η Επίτροπος. Ουσιαστικά μπαίνουμε στο τρίτο τμήμα ε, τη σημερινή συζήτηση. Τι μέτρα δηλαδή μπορούν και πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του χάσματο αμοιβέ ανδρών και γυναικών. Χαίρομαι πάρα πολύ Καλωσορίζω την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Αρμόδιο για Δικαιοσύνη, Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια, την κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ. Θα σας δώσω, αν είστε έτοιμοι, το λόγο ευθύς αμέσως. I'm always ready when... Πάντα έτοιμη είμαι όταν με ρωτάτε, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω τόσο πολλοί αριθμούς εδώ. Αυτό καταδεικνύει ότι πολύ καλά εξέλιξε το θέμα της σήμερα το Κοινοβούλιο για να το συζητήσει με πολλούς άντρες και γυναίκες. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία, όπως ξέρετε, δείχνουν ότι τώρα είμαστε στο 16,4% της διαφοράς του μισθού άνδρων και γυναικών. Αυτό είναι μία μείωση σχετικά με το περσινό έτος που ήταν 17% αλλά νομίζω ότι δεν είναι και κανένας ιδιαίτερα ενθουσιώδης για το ρυθμό της μείωσης. Γιατί φέρεται ότι είναι πολύ αργή η ένταξη περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασία και η μείωση του μισθολογικού κενού προχωράει επίσης πολύ αργά βλέπουμε ότι παρόλο που υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και καμιά φορά τα αριθμητικά στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε ένα σφάλμα εκτίμησης γιατί υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν πολύ χαμηλό ε, μισολογικό χάσμα και αυτό οφείλεται μέλη στο γεγονός ότι πολύ λίγες γυναίκες εργάζονται. και οι περισσότερες εργάζονται σε ε, θέσεις υψηλού επίπεδου που δεν είναι πραγματικά τόσο μεγάλο το δασμολογικό αυτό χάσμα. Αυτό που βλέπουμε όμως ότι τελικά το πρόβλημα πλήττει όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Από τότε που υπάρχει η κρίση, διαβάσαμε ότι υπήρχαν ίσως πιο ανεδικέ επιπτώσεις για τους άνδρες στην αγορά ε, απασχόλησης. Ίσως είναι αλήθεια αυτό. Αλλά παρόλα αυτά οι γυναίκες επειδή εκ νέας αρχής σε χειρότερη θέση εξακολουθούν να βρίσκονται σε χειρότερη θέση από τους άνδρες και για την είσοδό τους στην αγορά απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Τα αριθμητικά στοιχεία από το 2010 καταδεικνύουν ένα κενό απασχόλησης 12% υπέρ των ανδρών. 70% είναι το ποσοστό για τους άνδρες και 60% το ποσοστό απασχόλησης για τους ε, γυναίκες σε στρογγυλούς αριθμούς. Αυτό το κενό των φύλων είναι ακόμα μεγαλύτερο όταν δούμε τα ποσοστά της ε, μερικής απασχόλησης γιατί ξέρετε ότι ένα σημαντικό τμήμα της διαφοράς στους μισθούς οφείλει στο γεγονός ότι πολλές ε, γυναίκες εργάζονται σε μερική απασχόληση 8% άνδρες, 31% γυναίκες και αυτό πάλι βέβαια έχει επιπτώσεις στις μισθολογικές διαφορές Σας το λέω και το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω συνεχώς και το είπα και στους υπουργούς εργασίας στην Ευρώπη του 2020 έχουμε προβλέψει 75% ποσοστό απασχόλησης σαν στόχο. Αυτός ο στόχος δεν θα επιτευχθεί ποτέ εάν δεν εργαστούν και οι γυναίκες. Είναι σαφές. Μόνο οι άντρες δεν μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο αυτό. Για να το πετύχουμε χρειαζόμαστε οι γυναίκες να αρχίσουν να εργάζονται σε όλα τα επίπεδα και σε ψηλότερα επίπεδα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος της στρατηγική του 2020. Γνωρίζουμε επίση ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερα προσόντα από τους άντρε. και όσο πάει και ακόμα περισσότερα. Ίσως θα ακούσετε με τη συζήτηση αυτή όσον αφορά τις ποσοστώσεις. Εγώ πάντα λέω ότι οι γυναίκες αποτελούν το 60% των ε, αποφύτων πανεπιστημίων. Υπάρχει δηλαδή αυτό το ταλέντο. Α, ευχαριστώ. Βλέπετε, οι κύριοι εξακολουθούν να είναι ευγενείς. So, nevertheless, I continue. Πάνω αυτά θα συνεχίσω. Λοιπόν, αυτές οι συζητήσεις για τις ποσοστώσεις με κάνουν να δίνω πάντα αυτό το αριθμικό στοιχείο, ότι δηλαδή 60% των αποφύτων των πανεπιστημίων είναι γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ταλέντο, ικανότητες. Αυτό όμως δεν μεταφράζεται σε καλύτερες θέσεις απασχόλησης και καλύτερους όρους εργασίας για τις γυναίκες. Λοιπόν, έχουμε διάφορα στοιχεία δικέ μας που δεν είναι σωστά. Δηλαδή, η ποιότητα, το ταλέντο, δεν είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας. Αν κοιτάξουμε πού προέρχονται οι διαφορές, Μπορούμε ευτυχώ να δούμε ότι το νομοθετικό μας έργο ήταν καρποφόρο. Γιατί ξέρετε, έχουμε την οδηγία του 2006 που αφορά την άμυση ε, διάκριση, δηλαδή ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Και όσο πάει έχουμε λιγότερες ε, περιπτώσεις άμεσης διάκρισης, ακριβώ σαν αποτέλεσμα της ε, λειτουργία στον νόμο μας. Γιατί υπάρχει πάντα τόσο ε, μεγάλο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το χάσμα αυτό δεν αφορά μόνο τον ίδιο μισθό για την Αυτή είναι μια αρχή που έχουμε από το 57 Έχουμε μια οδηγία, εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη αυτή και στο 2013 θα υποβάλουμε μια ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της εν λόγω οδηγίας στην πράξη. Αλλά φαίνεται ότι ήταν πραγματικά καρποφόρα. Λοιπόν, δεν είναι η νομοθεσία και η ανεπαρχή της εφαρμογή που οδηγεί σε αυτό το τεράστιο μισθολογικό χάσμα. Άλλοι λόγοι υπάρχουν, πολλαπλοί. Αυτό που ανέφερα, το μεγάλο ποσοστό μερικής απασχόλησης, η αδιαμητρότητα, η γονική άδεια που παίρνουν οι γυναίκες πολύ περισσότερο από ότι οι και επίσης η συστηματική ανεπαρκής εκτίμηση των προσόντων των γυναικών που πιστεύω ότι αυτό είναι ένα οικονομικό σφάλμα, γιατί αν περισσότερες από τις ικανότητες αυτές χρησιμοποιούνται καρμοφόρα θα υπάρχουν λιγότερα οικονομικά προβλήματα, όπως απεδείχθη και στις πιο πρόσφατες ε, επιστημονικές έρευνες. Και επίσης οι γυναίκες είναι μαζικά παρούσες σε εκείνους τους τομείς που οι μισθοί ούτως άλλως είναι χαμηλότεροι. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μία πολύ, πολύ μορφή προσέγγιση αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα του μισθολογικού χάσματος. Θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν. Ξέρετε ότι αποφασίσαμε ε, να υπάρχει μία ενημερωτική εκστρατεία πριν από τρία χρόνια με στόχο να γίνει καλύτερη κατανόηση αυτών. Ξέρετε επίσης ότι υπάρχει αυτό το δίκτυο των εταίρων της εκστρατείας. Πολλοί από αυτούς φαντάζομαι είναι εδώ σήμερα και πολλές φορές αυτοί ε, μεταβιβάζουν και διαδίδουν τα μηνύματα της εκστρατείας. Υπάρχει μια στρατηγική ενημέρωση προς τους εργοδότες και εργαζομένους όσον αφορά την, τον ίδιο μισθό για την ίδια εργασία. Υπάρχει επίσης η Ευρωπαϊκή η μέρα της ίσης αμοιβή 2 Μαρτίου. Καλύτερα από πέρσι, οπότε στις 4 Μαρτίου. Μια μικρή πρόοδος δηλαδή. Αυτή είναι η μέρα κάθε χρόνο που αναλογεί στις ε, περισσότερες μέρες που πρέπει να εργαστεί μια γυναίκα στην Ευρώπη για να έχει τον δύο τον ίδιο μισθό. Τρεις, τρεις μέρες κερδίσαμε. Πρόοδος για αυτή. Όχι μεγάλη, αλλά πρόοδος. Η Κομισιόν προετοίμασε ένα web clip που καταδεικνύει το παράλογο του ε, μισθολογικού αυτού χάσματος βάση του φίλου. Θα ήθελα να σας πω να το δείτε και να το διαδώσετε κιόλα. Θα το δούμε. Α, πολύ ωραία. Α, θα το δούμε σε λίγο. Ωραία. Ξέρετε, ότι οι εργοδότες είναι οι κύριοι παίκτες για την αντιμετώπιση του μισθολογικού αυτού χάσματος. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αυξηθεί η γνώση για το κενό αυτό. Προετοιμάσαμε ένα σχέδιο πρόσφατα, ακριβώς με αυτό το στόχο, που θα βοηθήσει οι εταιρείε να κατανοήσουν καλύτερα αυτό το κενό, τις αιτίες, τις επιπτώσεις και να μπορέσουν να υποστηριχθούν εκείνες οι εταιρείε οι οποίες θέλουν να προωθήσουν την ισότητα στον τόπο εργασίας. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της εργασίας μου για τις ποσοστώσεις είδα πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει πάντα μια εξήγηση βασιζόμενη στην στο επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν περισσότερες γυναίκες σε όλα τα επίπεδα, δεν επιβαρύνει μια εταιρεία, αλλά την βοηθάει να αυξήσει τα έσοδά της. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε συνεχώς, συνεχώς σαν μάντρα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ε, βοηθήσουμε τις γυναίκες. Επίσης οι εθνικές αρχές είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, στις ε, προσπάθειες αυτές. Χρειάζεται να ενθαρρύνονται σε επιχειρήσεις, οργανώσεις επιχειρήσεων, ε, τους κοινωνικούς εταίρους, τα εμπορικά επιμελητήρια κλπ. κλπ. Χαιρετίζω τις δράσεις κάποιων κρατών μελών όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα. Ορισμένου ξέρουν το LOGIP, παραδείγματος που πρώτα χρησιμοποιήθηκε στην Ελβετία και τώρα στη Γερμανία που ε, διευκολύνει τις ε, εταιρείε να αναλύσουν τους λόγους για το μισθολογικό κενό και να τους βοηθήσουν να το μειώσουν. Η Κομισιόν ενθαρρύνει αυτές τις δράσεις και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την βοήθεια που μας προσέφερε και Ιδίω την κυρία Μπάουερ με την έκθεσή τη για το μισθολογικό χάσμα. Θα εργαστούμε μαζί σας πάνω σε αυτή σας την έκθεση που προωθείτε τώρα και θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε. Θα κάνω ό,τι μπορώ και εγώ και ό,τι μπορώ να πείσω τους συναδέλφους από την Κομισιόν να το κάνουν γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε αυτή την ανομαλία στις κοινωνίες μας. Σας ευχαριστώ που μας βοηθείτε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Thank uh, Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρέντινγκ. Χαίρομαι πολύ που καταφέρατε να βρείτε χρόνο να, ήρθε, να έρθετε εδώ σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Να δούμε και ένα βιντεάκι τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. It's really good, I think. <laughs> Νομίζω είναι πολύ καλό, ε. Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, τώρα και ξεκινάει με το γύρο έρωτα απαντήσεων, ε, κυρίως προς την κυρία Ρέντινγκ που πρέπει σύντομα να μας εγκαταλείψει. Τέσσερις είναι οι ομιλητές. υπενθυμίσω ότι 24 Απριλίου στην Επιτροπή της συνεδρίασης, ε, στη συνεδρία της Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας θα είναι η κυρία Ρέντινγκ, άρα να το έχετε υπόψη σαν ε, παρακαλώ εκπρόσωπος της Κυπριακής Βουλής. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα κάθε επιτυχία σε όλες ε, τις γυναίκες, τόσο τις παρούσες όσο και τις απούσες, ε, που τους εύχομαι χρόνια πολλά για την Παγκόσμια Μέρα Γυναικών, ε, υγεία, ευημερία, πρόοδο. Εύχομαι. Με πολύ μεγάλη χαρά απευθύνομαι στην συνεδρίασή σας που έχει ένα τόσο σημαντικό θέμα. Στη δική μας χώρα, Υπουργό Κοινωνικών ε, Θεμάτων εφαρμόζει ένα πρόγραμμα που θα ολοκληρωθεί το 2015 δράσεις για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος και συγχρηματοδοτείται το πρόγραμμα αυτό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που απαρτίζεται από ένα μείγμα πολύ καινοτόμων μέτρων. Μεταξύ αυτών είναι η εκπαίδευση και ο έλεγχος ε, της εφαρμογής ε, των ίσων ε, της ίσης αμοιβή και στην πρωτογενή νομοθεσία. Θα γίνουν επίσης ε, επισκέψεις μελέτης από τους επιθεωρητές σε άλλες χώρες για να εξοικειωθούν με τις τεχνικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Επίσης, Συγγνώμη σας διακόπτω, λέει ο Πρόεδρος, αλλά έχετε ερωτήσεις προς την κυρία Ρέντινγκ. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένα να στηρίξουν το πρόγραμμα της χώρας μου αλλά και άλλων χωρών για να έχουμε μεγαλύτερη ισότητα και στις αμοιβέ αλλά και σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ποια είναι τα προγράμματα της Επιτροπής αντιπρόεδρος της οποίας είναι και η κυρία Ρέντινγκ. Σα Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Περνάμε στον επόμενο μιλητή. Από την Ελληνική Βουλή, κυρία Ελένη, έχετε το λόγο για πάνω δύο λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να κάνω κάποια ερώτηση. Αν θέλετε μπορώ να περιμένω να τοποθετηθώ στο τέλος ε, στα δύο λεπτά που μου αναλογούν αφού ολοκληρωθεί. Όχι, συνεχίστε. Ευχαριστώ. Στη χώρα μου η δομή της ελληνικής οικογένειας... Μπορείτε να παρέμβετε ε, και μετά αν θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά την κυρία Ρέντινγκ. Αφήσουμε το χρόνο στην ε, κυρία Επίτροπο να ολοκληρώσει και στη συνέχεια θα τοποθετηθώ. Ωραία. Θα σας δώσω πρώτα το λόγο. Πρώτα σε εσά, σας το υπόσχομαι. Οπότε να δώσω τον λόγο στην κυρία Μεντέρ από την Πρωτογαλία. Αλλά επαναλαμβάνω, αν μόνο έχει να υποβάλει το ερώτημα στην κυρία Ρέντινγκ. Ε, ε, Λυπούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχα ετοιμάσει μία παρέμβαση σύντομη, αλλά έχω και ένα ερώτημα προς την κυρία Ρέντινγκ. Α θέσω το ερώτημά μου, χωρίς την παρέμβαση. Βέβαια, ε, είναι λίγο άστοχο, είναι λίγο κενό το, το ερώτημα αν δεν έχει προηγηθεί παρέμβαση. Οπότε ή θα μιλήσω αφού φύγει η κυρία Ρέντινγκ. Να εξηγήσω κάτι, λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Ρέντινγκ το αργότερο στις 12 πρέπει να φύγει. Γι' αυτό θέλω να δώσω έμφαση τώρα στα ερωτήματα προς αυτήν, γιατί αν τα θέσετε απουσία της δεν θα μπορεί να απαντήσει. Ναι, αλλά πόσο χρόνο μου δίνετε κύριε Πρόεδρε. μπορείτε να λάβετε το λόγο μετά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν έχετε ερώτηση, μπορείτε να την κάνετε τότε. Οκ, okay, τότε θα μιλήσω μετά. Ευχαριστώ. Mrs. Ε, Kochmerin. Η κυρία Κοχμερίν, πώς είναι το λόγο, για προβλεφτή. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα έχουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, η μισθό για την ίδια εργασία. Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτό. Και βέβαια νομίζω ότι αυτό το ερώτημα θα πρέπει να λυθεί επιτόπου. Δηλαδή κάποιος που εργάζεται καλά θα πρέπει να αμείβεται και καλά. Αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι φαίνεται η αγορά δεν λειτουργεί προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό σίγουρα σχετίζεται και με το γεγονός ότι υπάρχουν εδώ διάφοροι παράμετροι, διάφορα στοιχεία τα οποία ίσως δεν περιμέναμε ότι θα έπαιζαν ρόλο στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό θα ήθελα να μου πει η κυρία Ρέντινγκ πώς βλέπει το θέμα της αξιολόγησης εργασίας στην Κομισιόν. Δηλαδή αν κανένα κάνει την ίδια εργασία ακριβώς. Ένας άντρας και μια γυναίκα κάνουν ακριβώς την ίδια εργασία και παίρνουν κάποια αμοιβή. Είναι πολύ εύκολο να δούμε ποια είναι η διαφορά. Αν έχουν δύο διαφορετικές απασχολήσεις ένας μηχανικός και μία νοσοκόμα παραδείγματος χάρη. Πώς ε, αξιολογείται εκεί η εργασία γιατί ο ένας παίρνει παραπάνω και ο άλλος ε, λιγότερα. Αυτό είναι θέμα της, αγο... αγοράς, αλλά αυτοί οι μηχανισμοί της αγοράς είναι βάσιμοι. Είναι πολύπλοκο το θέμα κατά τη γνώμη μου, γιατί παίζουν βέβαια και πολλοί κοινωνικοί ε, παράγοντες. Εμείς τι θεωρούμε σαν κοινωνία σημαντικό, αξιόλογο, και θεωρεί η Κομισιόν ότι εκεί πρέπει να δράσουμε, μπορούμε να δράσουμε κλπ. Και τέλος θα ήθελα να σας συγχαρώ για την αποφασιστικότητά σας να εξετάσετε ένα θέμα, το σας, που είναι τόσο α, φιλεγόμενο, τόσο αντιφατικό, αλλά όλα αυτά συνεχίζετε να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό θα να σας συγχαρώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σονισεβά έχει το λόγο του Ευρωπαϊκού Εκνοβούλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να χαιρετήσω και εγώ την παρουσία και την έκθεση της ε, Αντιπροέδρου Ρέντινγκ για τη θέση των γυναικών ε, στα, οικονομικά, στα όργανα οικονομικών αποφάσεων. Λέτε ότι πόρο απέχει του να είναι πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ισότητα ανθρώπων και γυναικών και έχω δύο ερωτήσει προς την Επίτροπο. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζω την απόφαση να μην προχωρήσετε άμεσα στην ε, υλοποίηση δεσμευτικών μέτρων, αλλά να προβείτε καταρχάς σε μια εκτεταμένη δημόσια διαβούλευση, οπότε αυτό θα επιτρέψει να εγκριθούν τα κατάλληλα μέτρα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια πιο συγκεκριμένη ιδέα για το χρονοδιάγραμμα που έχετε ορίσει ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσει αυτέ κυρία Ρέντινγκ, και αποτελέσματα προσδοκάτε. Δεύτερο ερώτημα, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε μια από τις ιδέες που συζητούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε κάθε κράτος μέλος έχουμε φορείς επιφορτισμένους με την πρόθεση και την εποπτεία της ίσης μεταχείρισης, ισότιμης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών. Κυρία Επίτροπε, η ενίσχυση της εντολής αυτών των οργανισμών και η επαρκή τους χρηματοδότηση καθώς και η εκχώρηση νομικών εξουσιών σε αυτούς τους οργανισμούς νομίζω ότι είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο ως μέτρο για να πετύχουμε το στόχο του ίσως μισθός για ίση εργασία. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, έχετε κάποιες πρωτοβουλίες να μας παρουσιάσετε για τον τομέα αυτό. Κύριε, Κύριε Μπράντερ, επίσης Ευρωβουλευτής. Σας ευχαριστώ. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. <coughs> Βλέπετε, εδώ είμαι. Λοιπόν, είπατε δικαίω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που οδηγούν στην μισθολογική ανισότητα. Και είπατε ότι από το 57 και μετά η ισότητα η μισθολογική έχει εδραιωθεί στη συνθήκη της Ρώμης, ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν, δηλαδή δεν χρειάζεται δηλαδή, να υπάρχουν νόμοι, αλλά η πρόκειται είναι εφαρμογή των νόμων που υπάρχουν. Είπατε εσείς για τις ποσοστώσεις δικαίως, ότι δυστυχώ ε, δεν έδρασαν από μόνες του οι επιχειρήσεις και γι' αυτό χρειαζόμαστε νέα νομοθετικά μέτρα. Όσον αφορά την ε, μισθολογική ανισότητα βλέπουμε ότι το θέμα δεν λειτουργεί το σύστημα. Χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργώντας ε, μεγαλύτερη διαφάνεια και βοηθώντας τις νομοθετική διαδικασία με κάποιε συλλογικέ προσφυγέ, παραδείγματο χάρη. Ε, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτως ώστε αυτό το δίκαιο που ισχύει από το 57 να πραγματοποιηθεί στην πράξη. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο κύριος αγγεί έχει ερώτηση προς την ε, Επίτροπο Ρέντινγκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο Ρέντινγκ, την αρμόδια για θέματα αυτά, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χαιρετήσω την κυρία Edith Power. Θα το κάνω στα ουγγρικά. Θα ήθελα να χαιρετήσω, όπως σας είπα, την ε, κυρία Μπάρκ και να σε και μια ερώτηση. Η κυρία Πάουρη είναι Ουγγαρέζα αλλά ζει στην Σλοβακία και το 1920 ήταν θύμα ενός ε, μιας απόφασης ε, που έπληξε 5 εκατομμύρια Ούγγρους ε, το 1920 και θα ήθελα να σας ρωτήσω κυρία Ρέντινγκ τι λέτε για το θέμα ότι μία γυναίκα 99 ετών Ουγγαρέζα στη Σλοβακία χάνει την υπηκότητά της. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Και δεύτερη ερώτηση. Στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης οι μισθολογικές διαφορές, ιδίω σε εκείνε οι εταιρείες οι οποίες προέρχονται από την Δυτική Ευρώπη, είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Γιατί αυτό είναι απορίας άξιων. Και οι ουγγρικές εταιρείες εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, οι εταιρείες όμως της Δυτικής Ευρώπης που επενδύουν σε εμά διατηρούνται μεγάλες δημιουργικές διαφορές. Και τελευταία θα μιλήσει στο γύρο αυτό η Επίτροπος Ρέντινγκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το τέλος και να πω πως δεν πιστεύω ότι θα πρέπει στη συζήτηση αυτή να μιλήσουμε για αντιπαραθέσεις μεταξύ κρατών μελών για ζητήματα μειοψηφίας. Ε, ως προς την κοινοτική νομοθεσία, έχουμε ήδη σχετική κοινοτική νομοθεσία και το 2013 πρόκειται να καταρτήσουμε έκθεση για τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσία αυτής στα διάφορα κρατημέλη και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της. Ήδη σα είπα, όχι όμως με επιστημονικό τρόπο, γιατί δεν έχουμε ακόμη τα επιστημονικά πορίσματα για τη σχετική έκθεση, πάντως ε, από μια πρώτη ανάλυση της κατάστασης διαπιστώνω ότι η σχετική κοινοτική νομοθεσία και εφαρμόζεται σωστά και αποφέρει καρπούς. Και οι μισθολογικές ανισότητες έχουν διτό λόγο. Ο πρώτος είναι ε, ο μεγάλος αριθμός των γυναικών σε μερική απασχόληση, σε θέση μερικής απασχόλησης, κάτι που αναπόφευκτα μειώνει τα εισοδήματα, το μισθό τους. Και ο δεύτερος λόγος είναι το γεγονός ότι οι πολλές γυναίκες απασχολούνται σε χαμηλά αμοιβόμενε θέσεις εργασίας. Ή από τη στιγμή που η γυναίκα αναλαμβάνει μια τέτοια εργασία πέφτει ο μισθός σε σχέση με το αντίστοιχο μισθό των ανδρών. Είναι κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη αυτή. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε εκστρατείες ενημέρωσης και αφύπνισης. Γιατί στόχος ενημερωτικής εκστρατείας είναι να Αφυπνήσει στα κράτη-μέλη και τα συνδικάτα, γιατί οι φεμινιστικές οργανώσεις, οι γενικές οργανώσεις στρέφονται στα συνδικάτα και τα συνδικάτα πιέζουν τις ενώσεις εργοδοτών. Και η ανάλυση γίνεται αναεταιρεία, αναεπιχείρηση. Και οι επιχειρήσεις εκείνες που στο εσωτερικό τους έχουν ένα δίκτυο για να βελτιώσουν τη θέση των γυναικών στην επιχείρηση, ε, επιβραβεύονται, στηρίζονται, βοηθούνται και αναδεικνύονται και προβάλλονται στον υπόλοιπο κόσμο ως υποδείγματα προς μίμηση και θετικά παραδείγματα. Πολλοί εργοδότες ε, έχουν ε, εγκαινιάσει ειδικά σχέδια με το θέμα αυτό και μπορείτε να λάβετε και τις τεχνικές πληροφορίες για αντίστοιχα σχέδια, ώστε να παροτρύνετε και τους δικούς σας εργοδότες να εστερνιστούν αντίστοιχα σχέδια. Ε, επίσης, οι χώρες που ασχολούνται με το θέμα αυτό έχουν και το γνωστό μηχανισμό διαφάνειας και μάλιστα θα συμβούλευα όσους έχουν επαφή με επιχειρήσεις στις πατρίδες τους να χρησιμοποιούν αυτό το μηχανισμό όλο και περισσότερο και να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα μέσα, το υφιστάμενο υλικό για να εξασφαλίσουν τέτοια διαφάνεια στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο μέλλον πάντως θα ήθελα ε, να αναδείξω σε μία εκστρατεία τις επιχειρήσεις με τις καλύτερες επιδόσεις γιατί ένας τρόπος να στιγματίσουμε τα προβλήματα είναι να τα δακτυλοδεικνύουμε και άλλο είναι να προβάλλουμε θετικά ε, παραδείγματα, υποδείγματα ε, επιχειρήσεων που προσπαθούν να επιλύσουν ακριβώς αυτά τα προβλήματα, ώστε να γίνουν ε, μοντέλο και παράδειγμα προς και για, υπόλοιπες, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα νομικά μέτρα, δεν υποβάλαμε από την αρχή κάποια νομικά μέτρα για δύο απλούστατους λόγους πριν να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διοργανώσει δημόσιες διαβουλεύσεις και να πραγματοποιήσει και μελέτη επιπτώσεων. Δεν μπορεί η, νομική, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομική πρόταση χωρίς να ε, έχει προηγουμένως ε, οργανώσει διαβουλεύσεις και μελέτη επιπτώσεων. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλές ε, δυνάμεις ε, στις κοινωνίες μας. Μερικές φορές ε, δρούν και αντιμαχόμενα και αντιφατικά, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και το φαινόμενο της συσπήρωσης των δυνάμεων πολλές φορές στις κοινωνίες μας προς το στόχο που μας ενδιαφέρει. Και μάλιστα οι σχολές επιχειρήσεων στην Ευρώπη έχουν συσπυρώσει τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν ένα κατάλογο, ένα πουλ με ονόματα γυναικών που ε, λόγω της ε, υψηλής τους παιδείας και λόγω της ε, πλούσης πείρας τους μπορούν να, να απασχοληθούν αμέσως. 3.500 ονόματα περιλαμβάνονται, γυναικών περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό. Και πολλές φορές ακούμε το επιχείρημα δεν υπάρχουν ε, γυναίκες ε, σε διοικητικά συμβούλια. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα επιχειρήματα να τα καταπολεμήσουμε γιατί υπάρχουν και θετικά επιχειρήματα όπου οι ίδιες οι δυνάμεις της κοινωνίας συσπηρώνουν τις δυνάμεις του, ανασκουμπώνονται για να μας βοηθήσουν. Θα πρέπει και εμείς να τις βοηθήσουμε και να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για συρρήκνωση αυτών των μισθολογικών διαφορών, κρατώντας αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξή μας και βοηθώντας και στηρίζοντας αυτούς που προβαίνουν σε μια πιο συγκεκριμένη και πολύ θετική ανάλυση. Θα ήθελα να πω στον Κύπριο βουλευτή ότι θα συναντήσω σήμερα το απόγευμα Υπουργό της Κύπρου και θα συζητήσω μαζί του αυτό το θέμα προκειμένου να περιλάβουμε στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και αυτό το ζήτημα, ώστε να, απο, να αποδειχθεί η Κυπριακή Προεδρία χρήσιμη όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ για τη συμμετοχή σας στη συνεδρία αυτή. Ξέρω ότι έχετε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και ανηλυμένες υποχρεώσεις, γι' αυτό θα μας αφήσετε, αλλά σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε. Ευχαριστώ. Τέσσερις ακόμη ομιλητές μας έχουν απομείνει στον κατάλογο που τους εξαναγκάσαμε προηγουμένως σε μια πολύ απότομη διακοπή. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη και το χρόνο μας και η κυρία Ρέντινγκ, όπως σας είπα, είχε στη διάθεσή της μόνο ένα ημίωρο για τη συνεδρία σε αυτή. Γι' αυτό ήθελα και να της δώσω την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις. Επανερχόμαστε λοιπόν στον κατάλογο των ομιλητών πριν περάσουμε στο τρίτο και τελευταίο πάνελ. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Ελένη Τσαούση από την Βουλή των Ελλήνων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στη χώρα μου η δομή της ελληνικής κοινωνίας βοηθά τις γυναίκες να ανταπεξέλθουν στους πολλαπλούς ρόλους τους. Υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον που ευνοεί τη γυναίκα που θέλει να κάνει καριέρα. Στην ανώτερη εκπαίδευση είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα και μια αναντιστοιχία σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης όπως και στην πολιτική η νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό κολλημένη σε παλιά στερεότυπα. Η ισότητα κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και ειδικότερα με ένα νόμο το 2010, τον οποίο είχα την τιμή να εισηγηθώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εναρμονίστηκε το εθνικό μας δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 54 του 2006, με την οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα ίσης αμοιβή για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας σε αυτό το νομοσχέδιο το σημαντικό κομμάτι ήταν ο ορισμός του συνηγόρου του πολίτη ως αρμόδιου φορέα για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στις συνθήκες και τους όρους εργασίας συμπεριλαμβανομένης της αμοιβή και στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σημαντικό επίσης κρίνεται το ειδικό σχήμα συνεργασίας μεταξύ του συνηγόρου του πολίτη και του σώματος επιθεώρησης εργασίας το οποίο με την καλύτερη αξιοποίηση δυναμικού ειδικών γνώσεων εμπειρίας και τεχνογνωσίας και μέσα από την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών θα ασκεί την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων από ανεξάρτητο φορέα όπως επιτάσσει η οδηγία είναι γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προοδευτικό σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Στην πράξη όμως αποδεικνύεται ανεπαρκές. Το χάσμα στις αμοιβέ είναι μεγάλο ακόμα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία και στην Ελλάδα καταγράφεται στο 22%. Οι γυναίκες σήμερα και οι νέοι στη χώρα μου πλήττονται πολύ περισσότερο φυσικά από την φοβερή οικονομική κρίση οι μισθοί έχουν πέσει τόσο χαμηλά που δεν υπάρχει περιθώριο και για περαιτέρω αδικίες. Επειδή όμως στην ιστορία του έθνους μας οι γυναίκες ήταν εκείνες που με τους αγώνες τους κάθε φορά συντελούσαν ώστε να αναγεννηθούμε από τις τάχτες μας, έτσι πιστεύω και σήμερα η ανάταξη της εθνικής μας οικονομίας θα έρθει πάλι μέσα από τη δημοκρατία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία και φυσικά μέσα από το δυναμισμό των Ελληνίδων. Ευχαριστώ. Okay, thank uh, Καλώς ευχαριστούμε. Το λόγο η κυρία Ινές από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, είχα προετοιμάσει μία ομιλία, δύο λεπτά λέει ο πρόεδρος. Είχα προετοιμάσει μία ομιλία και για τις ε, Τρει ε, ομιλητρίε του τρίτου πάνελ, όχι μόνο για την κυρία Ρέντινγκ. Ε, θα ήθελα να τη διαβάσω τώρα και μάλιστα στα πορτογαλικά μου επιτρέπετε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αυτό που χαρακτηρίζει το θέμα της μη διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένα εγκάρσιο θέμα και καλύπτει, αγγίζει όλους τους κλάδους της κοινωνίας και τους τομείς. Βέβαια η διάκριση ξεκινάει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό και ακριβώς γι' αυτό συμβάλλει στην δυσκολία ε, ξεπεράσματος της διαφοράς μεταξύ των νομοθετικών κειμένων που πολλές φορές προβλέπουν σημαντικά ηχέγγυα και είναι πολύ προχωρημένη αλλά ε, δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ε, αδικία αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα με έναν με μια μεταρρυθμίση των ε, πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικών, εκπαιδευτικής πολιτικής και θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων και στόχων μας. Ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης δεν μπορούμε να μιλάμε για πολιτικές απασχόλησης και εργασιακές συνθήκες ή για εκπαιδευτικές πολιτικές αν ξεκινούμε από την αφετηρία ότι η πολιτικές αυτές θα πρέπει να, να εφαρμόζονται με ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και να μην δημιουργούν αδικίες. Όπως αναφέρθηκε πολύ σωστά, αν από νομοθετική άποψη θα πρέπει να μπορούμε να προσαρμόζουμε την νομοθεσία μας ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην έμπρακτη εφαρμογή. Για παράδειγμα, οι ποσοστώσεις είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, παρόλο που δεν είναι και πολύ αντικειμενικό. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα παιδαγωγικό μα έργο ώστε να προβούμε σε μια αλλαγή τη νοοτροπίας και των ανδρών και των γυναικών. Ιδιαίτερα που σε μερικού τομεί έχουμε παλινδρομήσεις και κοινωνικο οικονομικέ εξαιτία τη κρίση, αλλά και οι ε, παναχωρήσεις στο, σε ό,τι αφορά την αδιαφορία που δείχνουν οι νέες γενιές ή την έλλειψη γνώσης για τις διακρίσεις που, ε, παρατηρούνται και στην ιδιωτική ζωή και στην επαγγελματική ζωή. Γιατί τα ίχνη αυτής της διάκρισης ε, μερικές φορές μένουν ε, ανεξίτηλα. Για παράδειγμα, ο μύθος ότι οι γυναίκες ε, δεν εργάζονται. Οι γυναίκες ανέκαθεν εργάζονταν, απλώς δεν αμείβονταν ή οι αποδοχές τους ήταν εξευθελιστικές. Ο μύθος λοιπόν ότι οι γυναίκες ε, δεν εργάζονται δημιουργεί μια πολύ περίπλοκη κατάσταση γιατί ακόμη και σήμερα η εργασία ε, των γυναικών εργάζεται ε, για... αντιμετωπίζεται για μερικούς ως επιλογή. Αυτό που είναι υποχρέωση για τον άντρα, δηλαδή να εργάζεται θεωρείται ως επιλογή για τη γυναίκα. Αυτό είναι λάθος. Δεν υπάρχει καλή προσαρμογή των ωραρίων εργασίας προκειμένου να μπορέσει η γυναίκα να συμφιλιώσει την οικογενειακή με την επαγγελματική τη ζωή. Επίσης ενοχοποιούμε πολλές φορές τις γυναίκες που επιλέγουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, που δίνουν έμφαση στον επαγγελματικό τους βίο. Είναι λοιπόν απαραίτητο όχι μόνο να αναγάγουμε αυτό το θέμα σε προτεραιότητα όλων των πολιτικών και των εθνικών και των κοινοτικών, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι με σημαντικές ενημερωτικές εκστρατείες, ε, ε, συστηματικές θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε μια αλλαγή της νοοτροπίας. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι εξή. Πώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να λάβουν υπόψη αυτά τα δύο στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για να εφαρμοστούν πολιτικέ εγκύτητε προ τον πολίτη και βιώσιμε, ιδιαίτερα στι χαλεπέ στιγμέ που διανύουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Uh, σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος και έχουμε και ακόμη δύο μιλητές. μιλήτρης συγκεκριμένα στο πάνελ. Ξέρω ότι πολύ θέλετε το λόγο, δυστυχώς όμως δεν μπορώ να σας δώσω το μικρόφωνο. Υπάρχει και ωράριο για τους διερμηνείς που θα πρέπει να αναπαυθούν, να διακόψουμε για, ένα, για το μεσημεριανό. Θα δώσω το λόγο στην Καταμάρα Βόντα για ένα μόνο λεπτό γιατί πρέπει να περάσουμε στο, περάσουμε στο επόμενο θέμα. Παρακαλώ, ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας. Želim predstaviti eh, en primer dobre prakse, relativno dobre prakse in to bom storila v manj kot dveh minutah. Hvala lepa. Θέλω να μιλήσω για μια καλή πρακτική, αλλά θα χρειαστώ πάνω από ένα λεπτό, γύρω στα τρία λεπτά. Το Σεπτέμβριο του 2010, 12 μόνο βουλευτίνες υπήρχαν ε, στη Βουλή. Τώρα το ποσοστό έχει πάει στο 30%. Έχουμε πλέον αποφασίσει Στι εκλογικέ λίστες ε, να είναι πολύ μεγαλύτερη η εκπροσώπηση των γυναικών. Το Σλοβενή Ποζιτίφ ήταν ε, το κόμμα με τις περισσότερες γυναικές συμμετοχές. Έχουμε λοιπόν ε, πολλές βουλευτίνες και βουλευτές βέβαια. συγκεκριμένα στην Επιτροπή Αναφορών. Η σύνθεση της Επιτροπής ε, για τα δικαιώματα των γυναικών ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εξέπληξε. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση ε, και των ανδρών είναι πολύ χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στα Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας μου, μία γυναίκα συγκεκριμένα και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. 4,4% είναι η διαφορά των αμοιβών των και γυναικών στη Σλοβενία. Δεν είναι πολύ κακό η υγιώς επίδοση, αλλά λόγω της κρίσης δυστυχώς έχουμε αυξανόμενα προβλήματα. Πια. Ο κύριος τώρα Μπαγής θα πάρει το λόγο, ο Τούρκος Υπουργός Ευρωπαϊκών Συγγνώμη Υποθέσεων, Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Είχα ε, δεχθεί την προηγούμενη εβδομάδα την κυρία Μπάουρ και την Επιτροπή της ε, με πολύ μεγάλη χαρά και τώρα χαίρομαι που βρίσκομαι στις Βρυξέλλες. Μπορεί να μην συμφωνώ απόλυτα μαζί της, αλλά η σιδερά κυρία της αγγλικής πολιτικής Μάργαρετ Θάτσερ είχε πει κάποια στιγμή αν θέλετε κάτι να υποθεί στην πολιτική ρωτήστε έναν άνδρα, αν θέλετε όμως κάτι να γίνει μια γυναίκα. Βλέπω σήμερα ότι οι γυναίκες ε, βουλευτές ε, στο Κοινοβούλιο έκαναν μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά για τη διοργάνωση ενός σημαντικού ε, συνεδρίου για τις ίσες αμοιβέ για ίση εργασία. Η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας πλέον κλείνει τα 35 της χρόνια. Εγώ θα έλεγα βέβαια ότι 365 μέρες το χρόνο θα έπρεπε να μας απασχολεί το θέμα της γυναικείας ισότητας, γιατί είναι και ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Είμαι ένα μέλος ε, πολιτικού κόμματος ε, στην Τουρκία που έχουμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια μέλη γυναίκες. Και νομίζω ότι και η επιτυχία του κόμματός μου ακριβώς από τη γυναικεία συνιστόσα προέρχεται. Και από την προσωπική μου εμπειρία μπορώ να σας πω ότι αν καταφέρετε να κινητοποιήσετε ε, αυτό το ποσοστό, το πολύ σημαντικό ποσοστό της κοινωνίας, θα σας εγγυηθεί και την απόλυτη επιτυχία. Να πω ότι στην Τουρκία είχαμε δώσει μετά την ε, καθιέρωση της Δημοκρατίας το 1923, είχαμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο πλαίσιο των προσπαθειών εξυγχρονισμού στα δικαιώματα των γυναικών. Η πρώτη γυναίκα διπλωμάτης ε, ορίστηκε το 1932. Έχουμε θέματα βέβαια με την ίση αμοιβή για ίση εργασία, ισάξια εργασία. Το βλέπουμε στην καθημερινή εργασιακή ζωή. Είμαι πολύ περήφανος γιατί στο Υπουργείο του οποίου ηγούμε έχουμε πάρα πολύ μεγάλη γυναική εκπροσώπηση. 58% των υπαλλήλων είναι γυναίκες και 65% ε, είναι γυναίκες στα ανώτερα κλιμάκια του Υπουργείου. Μου βλέπετε λοιπόν ότι ε, συνεχίζουμε παρά τις δυσκολίες ε, αυτές τις προσπάθειες, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στις ενταξιακές μας διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει πάντως να παραδεχτώ ότι η διαδικασία διαπραγμάτευση Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαδικασία μεταρρύθμιση που έχει κάνει την Τουρκία πολύ πιο δημοκρατική, διαφανή και με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, υπήρξε μια διαδικασία που δεν αφορούσε ε, μόνο τον άντρα, αλλά και τη γυναίκα στην Τουρκία. Όσο περισσότερε μεταρρυθμίσει κάνουμε, τόσο καλύτερο είναι και το βιωτικό επίπεδο, το επίπεδο διαβίωση και των γυναικών. Η διαδικασία λοιπόν μεταρρυθμίσεων ε, έτυχε στήριξη απόλυτη και του κυβερνώντο κόμματο αλλά και των κομμάτων τη αντιπολίτευση στην Τουρκία και έχει βελτιώσει το επίπεδο διαβίωση των γυναικών και στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή. Και δεν νομίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για να ασκηθεί βία από έναν άνθρωπο σε έναν άλλον. Και ακόμα χειρότερο αν το θύμα της βίας είναι η γυναίκα, είναι μια γυναίκα. Είναι σημαντικό αυτό, πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο για όλες τις χώρες και για κάποιες από τις πιο ε, στέρεες δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα θέματα όλοι μαζί. Και δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της ε, χάραξης ε, κάποιων δρόμων που έχουν να κάνουν ε, με προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή λόγω της θρησκείας, της καταγωγής κτλ. Είναι γενικότερο, είναι ευρύτερο το θέμα και η ισότητα ε, είναι γενικό ζήτημα και το θέμα της ίσης αμοιβή. Χαίρομαι που η χώρα μου τα τελευταία 9,5 χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά βήματα υπό την ηγεσία του Ερτογάν για την πρόθεση των θεμάτων των γυναικών και νομίζω ότι το εργατικό δυναμικό χρειάζεται γυναικείο εργατικό ε, δυναμικό και θα πρέπει πάνω σε αυτό να δουλέψουμε. Πρέπει να αναπτύξουμε ε, τις προσπάθειες αυτές την περαιτέρω. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Thank you very much for... Uh, Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ Μπαγή, για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση. Έχω κάποιες σύντομες ερωτήσεις που θα σας υποβάλει η κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχουμε υπουργό από υποψήφια χώρα στο πάνελ αυτό. Είναι σαφέστατο και χειρό μήνυμα ότι τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν προτεραιότητα και στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις επειδή είμαι ε, εισηγήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, ενώ των διαπραγματεύσεων για την διεύρυνση, σα συγχαίρω για τη νέα τουρκική νομοθεσία σε ό,τι αφορά ε, την πάταξη τη βία κατά των γυναικών, που όσο μιλάμε, κατά πάσα πιθανότητα εγκρίνεται στην Τουρκική Βουλή. Θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Γιατί για να λύσουμε προβλήματα όπω ε, μισθολογικέ διαφορέ, χρειαζόμαστε ένα ασφαλέ περιβάλλον για τι γυναίκε, χρειαζόμαστε ένα καλό εκπαιδευτικό σύστημα και φυσικά και μια εύρυθμη αγορά εργασία. Η συμμετοχή των γυναικών στην ε, αγορά εργασία ε, έχει αυξηθεί, έχει φτάσει στο 30% σήμερα και πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξηθεί περισσότερο. Αυτή είναι η φιλοδοξία και στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020. Θα μπορούσε ο Υπουργό να μα πει λίγα λόγια για το τι προσπάθειε γίνονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία, προκειμένου να ε, υλοποιήσει ίσω και του στόχου τη στρατηγική του 2020 η Τουρκία. Δεύτερη ερώτηση αφορά την, ε, τις διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο 19 στη, στις διαπραγματεύσεις είναι πολύ σημαντικό αυτό το κεφάλαιο γιατί αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Είναι σημαντικό εκτός από το κεφάλαιο 19 να εγκαινιαστούν οι συζητήσεις για το κεφάλαιο 23 που μιλά για τα θεμελιώδη δικαιώματα γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών. Σας ευχαριστώ κυρία Μποσκούρτ και σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ σημαντική έκθεση που καταρτήσατε που πραγματικά μας δίνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, επιλύει κάποια τωρινά προβλήματα και μας, αποτρέ... μας προφυλάσσει και από μελλοντικές, από δυσκολίες. Το 2011 πάνω από 8 εκατομμύρια γυναίκες απασχολούνται, απασχολ... βρήκαν μια δουλειά στην Τουρκία. Και αν το συγκρίνουμε το παρελθόν, το 2004 διαπιστώνουμε ότι ε, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ήταν 23,3%. Το 2011 αυξήθηκε στο 28,3% και ο στόχος μας για το 2023 όχι το 2020. Για το 2023 θα έχουμε την εκατοστή ε, πέτειο της σύγχρονης τουρκικής δημοκρατίας. Είναι να φτάσουμε στο 35% ε, συμμετοχή στον γυναικό στο εργατικό δυναμικό. Στο δικό μου Υπουργείο είναι 58% όπως σας είπα το ποσοστό απασχόλησης γυναικών. Και μάλιστα τα τελευταία 9,5 χρόνια πραγματοποιήσαμε πολύ σημαντικά βήματα προκειμένου να εστενιστούμε το κοινοτικό και εκτιμένο για την ισότητα των ευκαιριών και την ισότητα των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, να ενισχύσουμε την συμμετοχή των γυναικών και στην ε, πολιτική. Στο, στο τουρκικό κοινοβούλιο έχουμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό στην ιστορία μας ε, γυναικών πολιτικών βουλευτίνων. Δεν είναι ίσω αρκετό, αλλά για να φτάσουμε το 50% που είναι επιθυμητό στόχο θα πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά. Αλλά όπω ξέρετε, κυρία Μποσκούρ, το κόμμα μα είναι πολύ αποφασισμένο και προσιλωμένο στο στόχο αυτό. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 19 των διαπραγματεύσεων, μέχρι στιγμή έχουν ε, ανοίξει 13 ε, από τα 23 από τα 33 κεφάλαια. Έχουμε ακόμη 20 κεφάλαια που πρέπει να ανοίξουν. Βέβαια, 17 από τα κεφάλαια αυτά είναι μπλοκαρισμένα για πολιτικού λόγου, είτε από τα κράτη-μέλη είτε από το Συμβούλιο. Τρία είναι τα εναπομείναντα κεφάλαια. Το ένα από αυτά είναι το κεφάλαιο για την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση, το κεφάλαιο 19 δηλαδή. Πρόσφατα συμφωνήσαμε για ένα νομοσχέδιο εργασίακή εργασιακής με τι μη κυβερνητικές οργανώσεις και με εκπροσώπους ε, των συνδικάτων και των εργοδοτών και υποβάλαμε το νομοσχέδιο στην Τουρκική Βουλή, στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ευελπιστούμε ότι ε, η έγκριση αυτή τη νομοθεσία ε, θα είναι αρκετή απόδειξη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και την επιτομόφωνη απόφαση των 27 χωρών προκειμένου να ανοίξουν οι διαπραγματεύσει για το κεφάλαιο 19. Και ελπίζω οι ευρωβουλευτέ που εκπροσωπούν τη συνείδηση της Ευρώπης να ασκήσουν πιέσει στα κράτη του για να σταματήσει αυτή η ανόητη πολιτική του μπλοκαρίσματο των κεφαλαίων και να ανοίξει ο δρόμο για τι διαπραγματεύτικέ διαδικασίε, τι ενταξιακές διαδικασίες διαπραγματεύσει της Τουρκίας που είναι σημαντικέ και για τι γυναίκε τη Τουρκία. Σα ευχαριστώ και περνάμε στην τελευταία ομιλήτρια του πάνελ μα, που είναι η κυρία Edith Bauer συνάδελφος ε, και μέλος της Επιτροπής ε, ε, Δικαιωμάτων της Γυναίκας και Ισότητας των Φύλων. Είναι η συντάκτρια της γνωμοδότησης για την εφαρμογή της αρχής ίσης αμοιβή για άνδρες και γυναίκες για ίδια εργασία ή για εισάξια εργασία παρόμοιας αξίας. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι και εγκεκριμένοι επισκέπτες, θα ήθελα νομίζω να σας πω ότι πιστεύουμε όλοι ότι θα πρέπει να κλείσουμε αυτό το χάσμα. Το θέμα είναι πώς. Η έννοια της έκθεσης ήταν πρωτοβουλία 10 νεαρών γυναικών ευρωβουλευτών που προ... συνέταξαν μία επιστολή και την έστειλαν στις 8 Μαρτίου 2010 στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητώντας να υπάρχει μία έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας ε, ίδιου μισθού για την ίδια εργασία. Σύμφωνα με το κανόνα 40, το άρθρο 42 που λέει ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από την Κομισιόν να υποβάλει μια πρόταση ε, νομοθετικής πράξης ή τροπολογίας νομοθετικής πράξης μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε νέα νομοθετική βάση, το άρθρο 157 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, όπως αναφέρθηκε αρκετές φορές κατά διάρκεια της συζήτησης, ήδη έχουμε την οδηγία από το 2006 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής και ίσης μεταχείρισης άνδρων και γυναικών στον τόπο απασχόληση, το λεγόμενο ρίκα, που ανεκατέστησε μια παλιά οδηγία του 1975 για την προσέγγιση των νόμων των κρατών μελών για την εφαρμογή του νόμου της ίσης πληρωμής για άνδρες και γυναίκες. Παρόλο που εφαρμόζεται η οδηγία ΡΙΚΑΣ και που οι ε, προθεσμοί για την ε, μεταφορά της στις εθνικές νομοθεσίες ήταν 2008 έχουν οι εμπειρογνώμες την εντύπωση ότι δεν αλλάζει τίποτα στην νομοθεσία των κρατών μελών και δεν έχουν ακόμα επιβληθεί παρά ελάχιστες κυρώσεις στους ε, εργοδότες που καταπατούν την αρχή αυτή. Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρθηκε, έχουμε μια συμμετοχή 16,16 ,16, μια διαφορά μάλλον 16,4%. Άλλες είναι 1,9% και στην Πολωνία με ενδιαφέρον άκουσα ότι ο Πολωνός συνάδελφος αναφέρθηκε τουλάχιστον 20% υψηλότερο κενό από εκείνο που αναφέρει στη Eurostat και το ίδιο για την ε, Τσεχή Δημοκρατία και την Αυστρία. Παρόλο που υπάρχει η νομοθεσία για την ίση αμοιβή εδώ 40 χρόνια. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά στοιχεία γιατί δεν έχουμε τα στοιχεία από την Ελλάδα και την Εστονία. Στην Ελλάδα ακούσαμε 20%. Μάλιστα ένα συνάδελφο χθε αναφέρθηκε σε 30% στην Εστονία. Λοιπόν, ο μέσο όρο θα ανέβει. Παρόλο που έχουμε κάποια ισχύουσα ε, νομοθεσία, αυτή φαίνεται δεν είναι πολύ αποτελεσματική. Ε, και οπωσδήποτε δεν ε, έχουμε ουτοπίε ότι αρκεί μόνο η νομοθεσία για να μεταπιστεί το θέμα, αλλά παρόλα αυτά έχουμε στοιχεία που λένε ότι μπορεί καλύτερα να εφαρμοστεί η νομοθεσία. Μια που το θέμα του μισθολογικού χάσματος είναι πολύμορφο και οι επιπτώσεις είναι πολύμορφες και οδηγούν μεταξύ άλλων και σε κοινωνικές και οικονομικές ε, ε, διαφορές. οι ανισορροπίες ε, βασίζονται και στα στερεότυπα, παραδείγματο χάρη την επιλογή της, ε, ε, του, της μορφής εργασίας, της ειδίκευσης και πρέπει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ίμιση των διαφορών δεν εξηγούνται παρόλα αυτά. Θεωρούνται ότι είναι διαφορές που οφείλουν σε ανειδικές διακρίσεις. Η στατιστική δείχνει όμως ότι η διαφορά αυτή, το χάσμα αυτό αυξάνεται με την ηλικία, λόγω της ε, διαφοράς της παιδείας. Και ιδίω ε, αυξάνεται μετά την πρώτη άδεια μητρότητας. Και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε μια σφαιρική και πολυεπίπεδη απάντηση. Θα πρέπει να συνδυάσουμε νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα. Η έκθεση που συζητήθηκε στην Επιτροπή Γυναικών και θα συζητηθεί και στην Ολομέλεια είχε σαν στόχο να αναχνεύσει εκείνους τους τομείς της νομοθεσίας που μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος. Μια που Κομισιόν έχει την υποχρέωση βάσει του άρθρου 32 της οδηγίας Τρίκας να αναθεωρήσει την οδηγία αυτή και αν χρειαστεί να υποβάλει τροπολογίες Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013, όπως αναφέρει και η κυρία Ρέντινγκ, καλούμε την Κομισιόν να αντιμετωπίσει αυτή τη ε, διάκριση και να καταστήσει πιο αποτελεσματική νομοθεσία για τη μείωση του, ε, του μεσολογικού και χάσματος. Ο ορισμός δεν θα πρέπει να καλύπτει μόνο ακάθαρτο ωραίο μισθό, αλλά να είναι πιο σφαιρική. Η ανάλυση και η διαφάνεια των αποτελεσμάτων είναι επίσης σημαντική, γιατί καταλαβαίνετε ότι ακόμα δεν έχουμε απόλυτα βάσιμα στατιστικά στοιχεία. Θα ήθελα να τονίσω ένα μερικό θέμα. Δηλαδή υποχρεωτικές τακτικές εξετάσεις των μισθών στο οποίο θα επάγονται τουλάχιστον ε, επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν 10% και πάνω γυναίκες εργαζόμενοι. Γιατί πολλές φορές η μισθολογική πολιτική γίνεται καλυμμένα και μυστικά. Η αξιολόγηση, η ταξινόμηση το, της απασχόλησης είναι επίσης σημαντική. Αναφέρθηκε το θέμα της ίσης αξίας. Ε, έχω τον εντύπωση αυτό το θέμα δεν έχει ακόμα πάρει μια ικανοποιητική απάντηση. Και κάτι επίσης αναφέρθηκε όσον αφορά σώματα ισότητας και ε, νομική ε, εξουσία για την ε, πρόθεση της ίσης αμοιβή για ίση εργασία ή προ... προσαγωγή των υποθέσεων αυτών στα δικαστήρια. Πιστεύουμε επίσης ότι ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει να ενδυναμωθεί γιατί η ευθύνη των συνδικάτων στον τομέα αυτό είναι απόλυτα δεδομένη. Η πρόληψη της ανετικής διάκρισης. Να γίνει δηλαδή πιο γνωστό και κατανοητό το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ε, πληροφορίες και κατευθύνες γραμμές για την πράξη, κάποια μέσα ηλεκτρονικά ίσως. Παραδείγματος χάνει τη δυνατότητα συλλογικών συμφωνιών σε τοπικό ή τομιακό επίπεδο. Και τελευταία λύση ίσως και κυρώσεις. Εμείς δεν θέλουμε βέβαια να δημιουργήσουμε συμπληρωματική γραφειοκρατία και να την επιβάλλουμε στην οικονομία, αλλά σε ορισμένα κράτη-μέλη χρησιμοποιείται η μέθοδος Logit για την εξέταση των αιτήσεων για τις δημόσιες αγορές. Γιατί να μην χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή σφαιρικότερα και για άλλα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ξέρουμε λοιπόν φυσικά ότι δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα μόνο με την νομοθεσία και μόνο μία σφαιρική και πολυεπίπεδη προσέγγιση θα βελτιώσει την κατάσταση και θα κλείσει το χάσμα που υπάρχει. Όλοι όμως έχουν ευθύνη γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Θα πρέπει να κηρύξω το πέρας της συνεδρίασης. Ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια στα σουηθικά όμως. Ε, ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα, παρόλο που κράτησε αρκετά το πρωινό. Μας έδωσε πραγματικά πολύ τροφή για συζήτηση. Ακούσαμε πολλές ε, μεστές και εύστοχε παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη, όλου όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση, τους ε, εμπειρογνώμονες μας, τα μέλη του πάνελ. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Το θέμα της ισότητας ενδιαφέρει πάρα πολλού. Δυστυχώς ε, χρειάστηκε να διακόψω πολλούς ομιλητές, να τους περιορίσω το χρόνο αγόρευση. και λυπούμε, λυπούμε ειλικρινά είναι κρίμα και ντροπή μερικέ φορέ να διακόπτουμε του ομιλητέ, αλλά είναι πολύ θετικό ότι το ζήτημα αυτό είναι ενδιαφέρον για πολλού. Απλώ ε, είναι δύσκολο με το λίγο χρόνο που έχουμε να ικανοποιήσουμε όλου όσου θέλουν να μιλήσουν. Αλλά τουλάχιστον φάνηκε το ζωηρό ενδιαφέρον που υπάρχει αυτό το θέμα. Μιλήσαμε για τι διακρίσει στην αγορά εργασία και πολλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτό. Και όπως είπε η κυρία Στάρκερ, δεν αρκούν τα ωραία λόγια, δεν αρκούν τα ευχολόγια. Χρειαζόμαστε απτά μέτρα, συγκρίσιμα και καταμετρήσιμα. Και θα πρέπει να δούμε και άλλους τομείς, όχι μόνο την αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δούμε και το θέμα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Και πρόσφατα κάποιος με ρώτησε Ποιος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για να μειώσουμε αυτές τις μισθολογικές διαφορές. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς ένα μόνο σημαντικό παράγοντα, αυτό που βαρύνει περισσότερο για τις μισθολογικές διαφορές. Πάντως, αν σκεφτώ ένα μόνο παράγοντα, νομίζω ότι μακροπρόθεσμα το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να έχουμε πιο γενικευμένη εφαρμογή της αγωνικής άδειας και να τη μοιράζονται εξίσου άνδρες και γυναίκες στην γονική άδεια. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια πλεονεκτήματα, γιατί μέχρι στιγμής οι γυναίκες είναι αυτές που έχουν τις, έχουν τις περισσότερες ασχολίες χωρίς αμοιβή. Και μάλιστα οι εργοδότες προτιμούν να προσλαμβάνουν άνδρες παρά γυναίκες, γιατί θεωρούν ότι οι γυναίκες θα πάρουν άδεια μητρότητας και θα εγκαταλείψουν τη θέση τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχουμε μια πιο δίκαιη και ισομερή κατανομή της γονικής ώστε να, μοιράζονται, να τη μοιράζονται εξίσου άνδρες και γυναίκες. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Ήταν πραγματικά αθρώη προσέλευση. Τους ευχαριστώ θερμα, θερμά όλους όσους έλαβαν το λόγο και όσους παρακολούθησαν τις συζητήσεις. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Και επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω και μια αντιπροσωπή από το Μπαχρέιν, που παρακολούθησε τη συζήτηση και χαίρομαι θερμά που μπόρεσε η αντιπροσωπεία από το Μπαχρέι να έρθει σήμερα και να παρακολουθήσει τη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστούμε, ελπίζω να ήταν χρήσιμη συζήτηση και για σας. Τέλος, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι και για τους εθνικούς βουλευτές αλλά και για τους ευρωβουλευτές προβλέπεται μια δεξίωση, ένα κοκτέιλ ε, στο δεύτερο όροφο, αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίασης. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι θερμά όλους. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο για σας το πρωινό. Ευχαριστώ.